Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. ότι υπάρχουν πολλοί που απουσιάζουν, πολλά διενά έδρανα. Κάποιες πολιτικές ομάδες δεν εκπροσωπούνται πλήρως. Τουλάχιστον ε, βλέπω έναν σοσιαλιστή και δημοκράτη στην αίθουσα εδώ μαζί με μένα. Καταρχάς όμως, προτού σας ε, παρουσιάσω τον παλιό μας φίλο τον Γεώργ, θα ήθελα να σας πω ότι η ε, Τζεραλτίν στα δεξιά μου θα συνταξιδοτηθεί και θα φύγει στα τέλη Οκτωβρίου. Τον Τζέραν τον γνωρίζουμε πολύ καλά στην Επιτροπή Μεταφορών και ήταν μέλος της πρώην Επιτροπής ε, ΡΕΤ. Είναι από το 1999 εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι ένας από τους παλιούς θεματοφύλακες όπως λέμε. Είναι ειδικευμένο στα θέματα αεροναυτιλίας και έχει συμμετάσχει επίσης και σε διάφορα νομοθετικά κείμενα που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές συνεδριάσεις, σε πάρα πολλές αποστολές και επισκέψεις. Έχει έχει ασχοληθεί με διάφορα θέματα στα πλαίσια της γραμματείας. Οτιδήποτε και να έχει κάνει πάντως το έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Ήταν πάντα πολύ διακριτικός. Ε, οι συμβουλές του, οι παρενέσεις του ήταν πάντα πολύτιμες. και όπως θα λέγαμε στον Ιωμένο Βασίλειο, πάντα καταφέρνει τελικά να πει σωστά, να εκφράσει σωστά αυτό το οποίο ήθελε τελικά να πει εξ αρχής ο πρόεδρος. Προτού, ε, μάλλον δεν υπάρχει καν πορτρέτο του εδώ πέρα, ούτε έχει καν δικό μου πορτρέτο όπως στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί κάτι τέτοιο δεν ήθιστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως, ήταν ένας πάρα πολύ καλός σύμβουλος σε όλα τα νέα μέλη της γραμματείας, οποτεδήποτε, οποτεδήποτε έφτανε ένας καινούριο στην γραμματεία, απευθυνόταν ουσιαστικά στον Τζέραρτ. Ήταν ο πραγματικός μέντοράς μας. Επομένω θα μας λείψει και με αυτή του την ιδιότητα. Μία από τις πολύ σημαντικές ικανότητες που ενδεχομένω να μην γνωρίζετε είναι ότι έχει γράψει πολλά άρθρα και λόγους για τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής και πρώην πρόεδροι θα σας πούν ότι έχουμε συγγράψει κάποια καταπληκτικά, καταπληκτικά άρθρα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουμε γράψει εμείς, δεν γνωρίζαμε τίποτα για τα άρθρα αυτά, έχουν γραφτεί από τον Τζέραρτ. Ήταν πάρα πολύ καλός λοιπόν στην ιδιότητά του αυτή. Ξέρω λοιπόν ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά, πάντως θα συνταξιοδοτηθεί και θέλω ειλικρινά να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια εξ ονόματος ε, όλων των μελών της Επιτροπής και των προηγούμενων προέδρων της Επιτροπής και από τα πρώην μέλη της Επιτροπής αυτής θα θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν. Ευχόμαστε καλή τύχη, καλή υγεία, καλή σύνταξη και θα χαρούμε πάρα πολύ να σε ξαναδούμε εδώ πέρα αν πραγματικά θέλεις να ξανέρθεις στην Επιτροπή μας. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα στην 38η αναδιατύπωση του σιδηροδρομικού πακέτου μπορείς να ξανάρθεις εδώ πέρα για να μας δεις. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι έχεις κάνει και πραγματικά σου εύχομαι μια ευτυχισμένη συνταξιοδότηση. Okay, another quick announcement. Μια άλλη σύντομη ανακοίνωση θα γίνει μια συνεδρίαση στις 10 Νοεμβρίου, 5η 10 Νοεμβρίου το πρωί, 9 με 11.30. Ο λόγος για τη συνεδρίαση αυτή είναι ότι θα έχουμε μια μερίδα για το περιβάλλον. Θα γίνει μια παρουσίαση της νέας έκθεσης του Οργανισμού για το Περιβάλλον, προκειμένου να δούμε ποια είναι τα συστήματα ταυτοποίησης της επίπτωσης των μεταφορών στο περιβάλλον και με τον Επίτροπο Έντιγκερ στη συνέχεια θα έχουμε μία συζήτηση. Σας παρακαλώ να δείξετε μια κάποια ήπια στάση. Θα μιλήσουμε για τις εκπομπές των θαλασσίων μεταφορών καθώς επίσης και για το ETS. 10 Νοεμβρίου 9 με 11.30 θα γίνει αυτή η συνεδρίαση. Με ιδιαίτερη χαρά τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω για μία ακόμη φορά τον πρώην συναδελφό μας Γεωργ Γιάρζεμπόφσκι ο οποίος είναι συντονιστής για τα λειτουργικά τμήματα ενέργειου χώρου, FAB. Είναι όμως και FAB επειδή είναι fabulous όπως λέμε στα αγγλικά, είναι καταπληκτικός. Προσβλέπουμε λοιπόν, George, να μας κάνεις μια παρουσίαση. Προβλέπουμε στην παρουσίασή σου, έχεις τον λόγο και στην συνέχεια, αφού ολοκληρώσει την παρουσίασή του ο θα γίνει μια συζήτηση και θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον κύριο Πίτερ Γκρίφιτς. Έχεις το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι του μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά για μένα να είμαι παρόν ενώπιον σα για να παρουσιάσω την τρίτη μου έκθεση. Ελπίζω την έχετε όλοι στα χέρια σα. Προετοιμάστηκε από τους ε, συνεργάτες μου για τα θέματα αυτά και επειδή χρειάζεται να μοιράσουμε το χρόνο μας, ο Πίτερ και εγώ, θα είμαστε πάρα πολύ σύντομοι και εχμηρή και θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον περιορισμένο μας χρόνο για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Καταρχήν, θέλω να σας πω ότι η διαδικασία της δημιουργίας των FAB, των λειτουργικών τμήματων ενέργειου χώρου, έχει σταθεί κάπως απογοητευτική. Θέλουμε να υπάρχουν εννέα FAB τα οποία θα δημιουργηθούν με την ε, Συμφωνία των Κρατών Μελών, αλλά πρέπει να αποφασίσουν ποιες χώρες θα αποφασίσουν. Δεν είναι <clears throat> ο τρόπος με τον οποίο θα το σχεδίαζε κανείς από την αρχή. Από τα κάτω από τις χώρες αυτές ξεκίνησαν. Αλλά ακόμα εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το βόρειο ευρωπαϊκό το, του, Δούναβη, της Κεντρικής Ευρώπης και του, της Ανατολικής Μεσογείου. Ακόμα χρειάζεται να υπάρξει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και επίσης μεταξύ των ε, ε, υπηρεσιών Εναρίων Ελεκτών για να μπορέσουν όλα αυτά να για να μπορέσουν όλα αυτά να γίνουν μέχρι το τέλος 2012 χρειαζόμαστε οι συμφωνίες να υπογραφούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα ότι στο τέλος του χρόνου θα προλάβουμε να τα έχουμε όλα αυτά. Αυτή ήταν η υπόσχεσή τους, θα πρέπει να τους ε, υποχρεώσουμε να τηρήσουν την υπόσχεσή τους, αλλά αυτό είναι κάπως απογοητευτικό. Για τα τέσσερα φάμπο που έχουν γίνει διακρατικές συμφωνίες, μόνο το Ιρλανδοβρετανικό και το Δανεζικό-Σουηδικό δουλεύει καλά και δίνουν παραδείγματα βελτίστων πρακτικών στην περίπτωση Δανίας και Σουηδίας δημιούργησε μια εταιρεία συμμετοχών που, στην οποία συμμετέχουν δύο πάροχοι υπηρεσιών πλοήγησης. Βρέθηκε λοιπόν μια λύση για να μπορέσουν να συνενωθούν δύο θεσμοί και να λειτουργήσουν από κοινού με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό είναι ένα πολύ καλά, καλό παράδειγμα βέλτιση των πρακτικών. Η Αγγλία και Δανία, Σουηδία λοιπόν έχουν συνεργαστεί πολύ καλά. Το ΦΑΠ της Κεντρικής Ευρώπης έχει υπογραφεί το Μάιο του 2011, αλλά ακόμα ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να οργανώσουν καλύτερα τη συνεργασία τους. Αυτό το οποίο δημιουργεί προβλήματα είναι το ΦΑΜΠΕΤ, το ΦΑΠ της, Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης. Είναι το σημαντικότερο γιατί καλύπτει περίπου 50% του ενάριου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει γίνει η υπογραφή το Δεκέμβριο του προηγούμενου χρόνου και το ΦΑΜΠΕΚ προχώρησε σε πολλές ε, συζητήσεις και συναντήσεις χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα γιατί οι υπάροχοι υπηρεσιών για απλοήγηση προσπαθούν να διατηρήσουν το εθνικό τους χώρο και το εθνικό τους εισόδημα και η εντύπωσή μου είναι ότι το εγχείρημα αυτό για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού ως ΦΑΜΠ γιατί αυτό είναι η ιδέα, να κάνουμε κάτι ως φαμπ όλοι μαζί. Αυτό ακόμα δεν τους έχει γίνει κατανοητό. Τα λέω λιγάκι έξω από τα δόντια, αλλά ο στόχος μου είναι να σταθώ ένας αντικειμενικός παρατηρητής της κατάστασης και να σας δώσω μια έκθεση για τα πεπραγμένα τους. <clears throat> Χρειάζεται μια πιο μεγάλη δέσμευση από τα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη θέλησαν από κάτω προς τα άνω να αυτοοργανωθεί το σύστημα αυτό. Δεν θέλανε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι είναι δική τους υποχρέωση να οργανώσουν τα FAB στα τρία απαραίτητα επίπεδα και όχι μονάχα σε επίπεδο διακρατικής συμφωνίας. Αυτό είναι δύσκολο. Έχει τεχνική κυριαρχία, μπορεί να γίνει κάτι με διεθνή συμφωνία, ρύθμιση αυτού του είδους. Αλλά πέραν αυτού του επίπεδου, του διακρατικού, πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά αυτοί οι φορεί. Και μην ξεχνάτε ότι δεν το κάνουμε αυτό για τυπικού λόγου. Το κάνουμε αυτό γιατί τα ΦΑΜ μπορούν να αυξήσουν την χωρητικότητα μεταφορά, να είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με το κόστο, να βελτιώσουν τη διαχείριση των, ε, των και φυσικά να αυξήσουν και την ασφάλεια στις χώρες μας και στις τρίτες χώρες που συμμετέχουν. Για να έχουμε λοιπόν μια πραγματική δέσμευση από τους Εθνικούς Υπουργούς Μεταφορών, θα ήταν χρήσιμο η Επιτροπή Μεταφορών να απευθυνθεί στο Συμβούλιο. Ξέρω ότι ήδη συζητήσατε μαζί με την Ουγγρική Προεδρία τον Ιούλιο και ίσως θα μπορούσατε και με την ε, τωρινή Πολωνική Προεδρία να το θέσετε το θέμα αυτό των ΦΑΜ, γιατί θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πολύ θετικό παράδειγμα η Πολωνία αν υπογράψουν το βαλτικό FAB γιατί εκεί πέρα είναι μάλλον εύκολο να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Και αν τα μέλη <clears throat> της Επιτροπής Μεταφορών εξετάσουν αυτή την ε, έκθεση και δούνε αυτά που περιέχονται για το ΦΑΜ της δικής τους χώρας, ίσως μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους εθνικούς υπουργούς τους, λέγοντας ότι το έχουμε συμφωνήσει όλοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για αυτή την νομοθεσία τι κάνετε για να την εφαρμόσετε στην πράξη. Γιατί θυμάστε αυτά που λέγαμε παλιά στο Κοινοβούλιο, κάνουμε πολύ καλή νομοθεσία, παράγουμε πολύ καλή νομοθεσία, αλλά αυτή έχει αξία μόνο αν εφαρμόζεται. Και αυτό είναι υπόθεση πολλές φορές των κρατών μελών. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί δεν θέλω να ενοχλήσω τον Μπράιαν και να του πω ότι πρέπει να επιτεθούμε και πάλι σε ένα εχθρικό στόχο. Έχουμε επίσης το οδικό χάρτη για, την, ε, για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο όπου ο εισηγητής έχει ζητήσει να υπάρξει μια συγχώνευση των εννέα προβλεπωμένων ΦΑΜ σε λιγότερα ΦΑΜ για να υπάρξει πραγματικά ένα πλεονέκτημα για ενιαίους ευρωπαϊκούς ε, εφέρες. Αλλά η υπάρχοι <clears throat> υπηρεσιών πλοήγησης στην Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο ήδη προχωρούν προσπαθώντας να εξασφαλίσουν και μία συγχώνευση των δύο ΦΑΠ σε ένα μονάχα. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα λοιπόν για να είναι βάση της έκθεσης του εισηγητού σας. Ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας. Είμαι έτοιμος να απαντήσω τα ερωτήματά σας και αν θέλετε μπορώ να πω περισσότερο και για τα μεμονωμένα FAB. Ευχαριστώ πολύ Γεώργ. Το πρώτο ερώτημα έρχεται από τον κύριο Γκρός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Γεώργ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την εργασία και την προετοιμασία σε αυτά τα θέματα και εμείς είμαστε φυσικά απογοητευμένοι όπως και εσύ για τα αποτελέσματα αυτό όμως Οφείλεται στη δική σου προσπάθεια κάθε αντίθετο. Δεν είναι εύκολο το έργο σου, κανένα ε, συντονιστή δεν έχει εύκολο στόχο, δεν έχει εύκολο εγχείρημα μπροστά του, αλλά θα έπρεπε να βρούμε τρόπο να καταλάβουμε γιατί προχωράν τα πράγματα τόσο αργά. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα FAB μειώνουν το κόστος, κάτι που θέλουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτουν σε αποδοτικότητα και περισσότερη αποδοτικότητα σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια, ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα όλους μας και επίσης όλα αυτά σημαίνουν και λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Λοιπόν, η επικοινωνία προς τα έξω θα πρέπει να τονίσει κατά την άποψή μου αυτές τις τρεις πτυχές ώστε η αντιμετώπιση των ΦΑ που φαίνεται πολύ τεχνικό θέμα να γίνει κάτι πιο ζωντανό και επικοινωνιακό προς τον έξω κόσμο. Και για μένα αυτά τα θέματα συνδέονται με τα δύο ερωτήματα που θέλω να θέσω Πρώτον, πώς βλέπει ο συντονιστής του ΦΑΜ το μέλλον, πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει, να συνεργαστεί, να παίξει κάποιο ρόλο για να προωθηθεί αυτό το συνολικό θέμα. Και το δεύτερο ερώτημα, εκεί όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά λόγω ε, πολιτι... έλψης πολιτικής θέλησης. Αλλά υπάρχουν ακόμα τεχνικά θέματα τα οποία ε, παραμένουν, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτά λοιπόν είναι τα ερωτήματα τα οποία εγώ θα ήθελα να θίξω γνωρίζοντας ότι εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες να δούμε ποια είναι η πιο πρόσφορη μορφή παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα τα πολιτικά κόμματα στο Κοινοβούλιο θεωρούν ότι όχι μόνο ήταν μια καλή πρόταση τα ΦΑΜ, αλλά ότι πρέπει εγκαίρως στο τέλος του πρώτου χρόνου για, αυτό, για την πρώτη φάση και οριστικά το, 2000, το 2012 θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρω. Ο κύριος Αλκαδραουή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γεζεμπόφσκι για την παρουσίαση που μας έκανε, αλλά και για το σαφές μήνυμά του, δηλαδή ότι τελικά δεν είναι και όλα ρόδινα και δεν, όλα, και δεν προχωρούν όλα με, όπως τα είχαμε προβλέψει. Πρέπει να σας πω ότι με εξέπληξε λιγάκι η, η όλη κατάσταση. Δηλαδή είναι εύκολο να υπογράφουμε, να συνάπτουμε συμφωνίες κτλ από εκεί και πέρα όμω τι γίνεται. Όλα αυτά πώς ε, μεταφράζονται σε πράξη. Και πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει και η Επιτροπή Μεταφορών να ασχοληθεί λίγο με το τι γίνεται σε κάθε χώρα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι και η πρώτη απόπειρα την οποία να ε, κάνουμε τώρα για να πετύχουμε τα, τους ενιαίους θέρες. Ε, ήδη έχει ξεκινήσει μια προσέγγιση και από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή ξεκινώντας από τα κράτη-μέλη, να τα αφήσαμε να προχωρήσουν. Από ό,τι φαίνεται όμως ακόμα δεν έχουμε καμία επιτυχία, εξού και διαρωτώ με μήπως θα έπρεπε να υιοθετήσουμε πιο αυστηρή νομοθεσία για να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. θα πρέπει σαν Επιτροπή Μεταφορών να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτά αποτελέσματα. Και συμφωνώ με αυτά που είπε ο Μάθιου προηγουμένως ότι υπάρχουν τεχνικά θέματα. Θέματα τα οποία σχετίζονται με την οργάνωση, ε, το καταστατικό για το προσωπικό. Αυτά αν επιληθούν, θα μπορούσαν να προχωρήσουν το όλο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις που να βρίσκουν σύμφωνους και όλους τους ενδιαφερόμενους. θα μπορούσαμε να δούμε, μήπως θα μπορούσαμε να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο με τον συνάδελφο Γεζεμπόφσκι, να συγκεντρώσουμε τους ενδιαφερμένους γύρω από ένα τραπέζι και να πιέσουμε για να πετύχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, για να ολοκληρώσω την ε, παρέμβασή μου, θα πρέπει και στην κοινή γνώμη να προβάλλουμε τη σημασία αυτού του θέματος, διότι μιλάμε για ασφάλεια, για αποτελεσματικότητα. Ακόμα και, και ε, οι στόχοι μας ε, για τις κλιματικές αλλαγές Νομίζω ότι οι ενιαίοι εθέρες θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά ε, τον περιορισμό των κλιματικών συνθήκων από ότι η ανταλλαγή εκπομπών. Κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ. Ε, ελέγχθη ότι πράγματι τα πράγματα αυτά δεν λειτουργούν. Ξέρω και καταλαβαίνω αυτή την απογοήτευση. Εγώ ξέρω ότι ο Γέργο είναι ένας άνθρωπος δυναμικός, ο οποίος καταφέρνει πάντα να πείσει όλους αυτούς οι οποίοι ε, τροχοπεδούν τις διαδικασίες. Αλλά αυτοί που δεν έχουν υπογράψει ακόμα τις συμφωνίες δεν τις έχουν υπογράψει. Θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ενισχύσουμε την ιδέα των ενιαίων ευρωπαϊκών εθέρων. Το ένα θέμα είναι να υπογράψουν τα κράτη-μέλη, αλλά το δεύτερο είναι να μπορέσει αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί κανεί, να το υλοποιήσει στην πράξη. Θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή με την Πολωνική Προεδρία. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να έχουμε μια μεγαλύτερη επιτυχία λόγω του Βαλτικού ε, ΦΑΠ και μετά θα έρθουν οι Δανείοι στην Προεδρία. Ξέρουμε ότι οι Δανείοι ω αυτοί που έχουν να δείξουν τι βέλτιτε πρακτικέ έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν το θέμα αυτό περισσότερο και ενδεχομένω να πείσουν του άλλου υπουργού μεταφορών και τα άλλα κρατημέρια στο Συμβούλιο για την ανάγκη να προωθήσουμε το, τα ΦΑΠ αυτά. Επομένως, το θέμα είναι να δούμε ποιος είναι αυτός με τον οποίο μπορούμε να έχουμε μια συνεργασία ποιο είναι αυτό ο οποίο διστάσει για να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούμε και κάτι άλλο το οποίο θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και εμείς φυσικά στις δικές μας εκλογικές περιφέρειες ενώπιον της κοινή γνώμης να κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε τον κόσμο, ίσως μιλώντας με αεροπορικές εταιρείες, με αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να έχουν πιο αποτελεσματικές και πιο αποδοτικές αεροπορικές μεταφορές, ώστε να μην εμπλέκονται μοναχά οι και οι υπουργοί, αλλά λιγάκι να αρχίσει και η κοινή γνώμη να ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. Ποια είναι η άποψή σου για αυτά λοιπόν, Γκέορ. E ευχαριστώ κύριε Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Γιαζεμπόφσκι, τον Γκέοργ, για την παρουσίασή του. Δεν είμαι απεσιόδοξη, αλλά δεν με εκπλήσει και η κατάσταση. Εάν ο Γκέαρκ δεν μπορεί να τους ταρακουνήσει, διαρωτώ με ποιος θα μπορούσε να το κάνει. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι όσο καλά όσο θα έπρεπε. Η νομοθεσία για τους ενιαίους εθέρες ε, είναι σε κρεμότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, θέλουμε και ζητάμε από τις αεροπορικές εταιρείες από τα αεροδρόμια να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή, γιατί ένα από τα βασικά θέματα είναι η συμφόρηση των εθέρων, ε, η μόλυνση, τα, οι τιμές των εισιτηρίων, ο ανταγωνισμός, εκτός από τα άλλα τα προφανή προβλήματα που αφορούν τη διαχείριση της αεροπορικής κυκλοφορίας. Και τα πράγματα δεν προχωρούν ε, τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Ε, δηλαδή θα πρέπει το 2012 να σκεφτόμαστε ότι θα αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα. Ε, λοιπόν, δεν, δεν υπάρχει ημερομηνία πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και αυτό το οποίο με απογοητεύει είναι ότι ε, ξέρουμε ότι εδώ υπάρχουν ε, συμφέροντα, ότι υπάρχουν ε, προβλήματα για κάποιες χώρες, πλεονεκτήματα, έχουμε ελεγκτές και κυκλοφορίας που είναι έμπειροι, αλλά που η, αυτό που τους ενδιαφέρει βασικά είναι η μισθή τους. Και εάν τα κράτη οι κυβερνήσεις δεν λαμβάνουν, λάβουν υπόψη αυτά τα συμφέροντα, τότε ε, ό,τι και να κάνει ο Γκέοργ δεν θα οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα. Και ούτω ή άλλως τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει, πρέπει κάτι να κάνουν. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο για να προχωρήσουν τα πράγματα όσον αφορά την διαχείριση των ε, εναέριων και ε, της εναέριας κυκλοφορίας. Άρα κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει όμως, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά ε, χαίρομαι ότι, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο η Ιρλανδία προχώρησαν, αλλά Υπάρχει μια έκθεση της Επιτροπής που δείχνει ότι πηγαίνουμε καλά, πηγαίναμε καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά τώρα σύμφωνα με την Κομισιόν το Ηνωμένο Βασίλειο έχει απορρίψει τα σχέδια ποια σχέδια είχαν υποβληθεί. Ήθελα να ακούσω ποια είναι η άποψη τη Επιτροπής και θα ήθελα, αν έχουμε χρόνο Πρόεδρε, να επανέλθω για να σχολιάσω αυτήν την απάντηση της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Τζόρτζ. Μην το παίρνει προσωπικά, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμεί. Μιλάμε για εμπορικές ε, εταιρείε, είτε είναι αεροπορικέ εταιρείε είτε είναι αεροδρόμια. Ξέρουν τι πρέπει να, κάνουμε, να κάνουν και ξέρουμε και εμείς τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να ασκήσουμε πιέσει και στις κυβερνήσεις και πρέπει να είναι μια συλλογική πίεση αυτή που ε, ασκείται. Και μετά αφού μίλησε ο κ. Γκρίφιθ θα επανέλθει, ο κ. Κόλουτσεκ. Πρέπει να σας πω, καταρχάς, ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώην συναδελφό μας, τον κύριο Γιαζεμπόφσκι και να τον διαβεβαιώσω ότι ασκώ μια πίεση ε, και εγώ με την σειρά μου ε, και θα συνεχίσω να ασκώ πιέσεις. Λοιπόν, για τα διάφορα ΦΑΜΠΑ. Ήδη στην ε, Τσεχία ήμουνα εισηγητής στο κοινοβούλιο μας για μια διεθνή συμφωνία για τις ε, εναέριες κυκλοφορία, για την εναέρια κυκλοφορία και τις εναέριες, εναέριες μεταφορές ε, όχι μεγάλων διαδρομών, μεσαίων διαδρομών. Έχω μια εμπειρία δηλαδή. Ε, ούτως ή άλλως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Εμείς Έχουμε στην Τσεχία ένα σύστημα διαχείρισης εναέρης κυκλοφορίας ιδιαίτερα σύγχρονο και πάντοτε είχαμε μια πολύ καλή ε, συνεργασία με την Σλοβακία. Ε, εκεί που υπάρχουν ε, προβλήματα είναι να συγκεντρώσουμε και τις, τους τέσσερις γύρω από ένα σημείο. Οι, οι Αυστριακοί θεωρούν ότι είναι τέλειοι. Οι Ούγγροι βέβαια δεν ήταν πάρα πολύ ε, καλή. Ήδη όμως στην Τσεχία στην δεκαετία του 30 του, στον 20ο αιώνα είχαμε, λέγαμε ότι ο αέρας είναι η θάλασσά μας. Το πρόβλημα είναι και τι θα κάνουμε και με την ε, Σερβία και το Μοντενέγκρο και το Ινθυρόμ τι θα γίνει με, την, με τον ενέργειο χώρο αυτών των, τριών, χωρών, των τριών χωρών. Επίσης, τι θα κάνουμε και με την Ισλανδία, που έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Και την Ισλανδία και την Γρυλανδία. Γιατί εκεί με τις χώρες αυτές έχουμε μια συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά την τι θα γίνει και με το νότιο κομμάτι της, ε, του Ατλαντικού. Επίσης, ε, τι γίνεται με το φάμπα Ευρώπης, ε, Κεντρικής Ευρώπης. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Κροατία και διαρωτώ με είναι κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε και εδώ. Εμείς σαν βουλευτές θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Το πρόβλημα είναι στην ε, κεντρική Ευρώπη, διότι είναι, πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν το ίδιο μέγεθος, ο καθένας θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι επικεφαλής και οι διαπραγματεύσεις ε, είναι δύσκολες. Κύριε Σφιντάντσα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Γερζεμπόφσκι για την ενημέρωση. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ και εγώ με τις ε, απορίες ε, και τις δυσκολίες που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Όλοι θεωρούμε ότι η ΦΑ, το ΦΑΜΠ είναι ένα, μια ψηφίδα πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση ε, των ενιαίων εθέρων και δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια συγκεκριμένη πρόοδος. Εγώ αναφέρομαι στο FAB Blue Med που είναι το πιο κριτικό αν θέλετε FAB ε, είναι και το πιο φιλόδοξο διότι έχουμε την φιλοδοξία να ε, ξεπεράσουμε ε, και την, τις ευρωπαϊκές χώρες και να συμπεριλάβουμε και ε, χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής. Έχουμε τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά έχουμε και τέσσερις χώρες της Μεσογείου που είναι συνδεδεμένες με διάφορα καταστώτα, παρατηρητές, αναπληρωτές κτλ. Εμείς έχουμε δει ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Καθυστέρηση η οποία επιδεινώνεται ε, λόγω ακριβώς της πολιτικής αστάθειας στις νότιες, ε, ε νότια όχθη της Μεσογείου μετά την ε, πολιτική άνοιξη του αραβικού κόσμου. Ε, το, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να αποφασίσουν οι τέσσερις χώρες της, ε, Ευρώπης και μετά να, να ε, εντάξουμε και τις άλλες τέσσερις χώρες στη συμφωνία αυτή. Πώς, εσείς, πώς το βλέπετε και ποιες είναι οι προθεσμίες που υπάρχουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη. Δεν είδα κανέναν άλλο να παίρνει το λόγο, επομένως θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, είναι ασυνήθιστο να συμφωνώ 100% και περισσότερο με την κυρία Φώστερ. Στην περίπτωση πάντως αυτή συμφωνώ 100% συν με την κυρία Φώστερ. Ενδεχομένως αυτό να έχει να κάνει με κάποιο δελτίο τύπου, δεν ξέρω. Πάντως έχει απόλυτο δίκιο στα όσα είπε σε σχέση με την επιβράδυνση αυτή την πολιτική βούληση, την απουσία πολιτικής, πολιτικής βούλησης. Εκεί έγκυται το πρόβλημα και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη αλλά και από τον κλάδο της βιομηχανίας να αρχίσουν να ακολουθούν ένα πολύ γρήγορο, γρηγορότερο ρυθμό. Και όντως η βιομηχανία μας δείχνει ότι θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς, ενώ εμείς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε μια ταχύτητα 747, τα κράτη-μέλη ακολουθούν ταχύτητα καμήλας. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε τώρα σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. Συμφωνώ λοιπόν με τα όσα είπε ο κύριος ε, Γιαρζεμπόφσκι. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε να επινοήσουμε προκειμένου να κάνουμε τα κράτη-μέλη να κινηθούν γρηγορότερα. Εκεί έγκυται το πρόβλημα. Αν δούμε το ΦΑΜΠΕΚ, το ΦΑΜΠΕΚ είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ΦΑΜΠ. Κατά την άποψή μου, το πρόβλημα εδώ πέρα είναι η έλλειψη βούλησης εξ ονόματος των κρατών μελών που απαρτίζουν το ΦΑΜΠΕΚ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ασκήσουν πίεση στα συνδικάτα των ε, ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας και δεν το κάνουν αυτό επειδή φοβούνται ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν απεργίες κτλ. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό έγκυται το πρόβλημα. Επομένως το πρόβλημα είναι πολιτικό. Θα περάσω τώρα και στα άλλα ζητήματα. Είμαι πεπισμένος απόλυτα ότι αν υπήρχε η απαραίτητη πολιτική βούληση στις χώρες που έχουν εντοπιστεί προβλήματα, δεν είχαμε την επιβράδυνση αυτή. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την πολιτική αεροπορία, δεν έχει να κάνει με τον ενέριο χώρο ή με κάποια αεροπορική εταιρεία, το πρόβλημα είναι πολιτικό. Ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη θάρρους, θα έλεγα, ορισμένων κυβερνήσεων προκειμένου να δώσουν απαραίτητη όθηση στο πρόγραμμα. Επομένως, ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Δανέζικη Προεδρία, λέει ο Πρόεδρος, προκειμένου να αποτελέσει μέρος της ημερήσιας διάταξής τους, των προτεραιοτήτων τους για την επόμενη Προεδρία. Δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο. παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια άτυπη συνεδρία των Υπουργών στην Δανία, στα πλαίσια της Δανικής Προεδρίας και θα ήθελα να με βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έτοιμά μου αυτό. Κατάλαβα τώρα τι είπαν τα κράτη-μέλη για κάποιε άλλε χώρε. Ο κύριο Κόλετσεκ και άλλοι συνάδελφοι μίλησαν. Και σαφώ ε, δεν ε, κάνουν λάθο. Πιστεύω όμως ότι είναι δύσκολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασκούμε πίεση στην Ισλανδία όταν δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώ μπορούμε να ασκούμε πίεση στο Μαυροβούνιο και στη Σερβία όταν δεν μπορούμε εμεί οι ίδιοι να ασκούμε πίεση στα κράτη-μέλη μα. Επομένω, ε, πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφεί για το τι κάνουμε και θα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο το ότι έχουμε την έκθεση αυτή από σένα, Γεώργ, και σε ευχαριστώ πολύ για την ειλικρίνειά σου, γιατί ήρθε εδώ και είπε τα πράγματα ξεκάθαρα. Δεν μα είπε ότι το, πρόβλημα θα τακτοποιηθεί, θα διευθετηθεί ε, μόνο του είπες ότι καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να γίνει πραγματικότητα, να ελοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό. Και καταβάλουμε προσπάθειες να δούμε δυσκολίες επειδή τα κράτη-μέλη δεν ανταποκρίνονται στις δικές τους υποχρεώσεις, στο τμήμα που τους αναλογεί. Σε ευχαριστώ πολύ και περιμένω να ακούσω τις απαντήσεις που έχεις να δώσει στα μέλη της Επιτροπής. Προσπαθώ να είμαι σύντομο και γιατί ξέρω ότι έχετε περιορισμένο χρόνο και ο Πίτερ πρέπει να αναφερθεί σε ένα άλλο θέμα. Δεν είναι θέμα τεχνικών προσκομμάτων. Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά δεν είναι τα σημαντικότερα. Το θέμα είναι και συμφωνώ απόλυτα ένα θέμα πολιτικής θέλησης από την πλευρά των αρμοδίων υπουργών. <clears throat> Κάποιοι υπουργοί δεν θέλουν ακόμα και να μιλήσουν μαζί μου, γιατί τότε θα πρέπει να πάρουν θέση για τα ΦΑΜ. Και δεν θέλουν να πάρουν καμία θέση για τα ΦΑΜ. Δεν του ενδιαφέρουν τα ΦΑΜ. Έχουν προβλήματα με φορτηγά, με σιδηροδρομικά συστήματα, με τα TNT, αλλά το FAB δεν βρίσκεται στην ατζέντα των Υπουργών. Επομένως πρέπει να το βάλει κανείς στην πολιτική ατζέντα των Υπουργών Μεταφορών. Τα πράγματα είναι έτσι γιατί. Και πώς θα κάνουμε κάποιες ε, βελτιώσεις. Εγώ δεν θα έφυγα καν αυτό το θέμα αν θέλουμε να λειτουργήσουν τα κέντρα εν αέριου ελέγχου από κοινού, αυτό δεν χρειάζεται καν να το κάνουμε στην αρχή. Αν θέλουμε να έχουμε εξοικονομήσεις και καλύτερη απόδοση, μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο. Άμα δείτε το προσωπικό των παρόχων υπηρεσίας για τα θέματα πλόγησης είτε στα Υπουργεία είτε σε εξωτερικές εταιρείες τουλάχιστον, 50% από τους εργαζόμενους είναι άτομα τα οποία παρέχουν απλώς υποστήριξη, δεν είναι ελεγκτές εν αερί. Είναι άτομα που κάνουν συστήματα υπολογιστών, εκπαιδεύουν τους ελεγκτές, ε, κάνουν αγορές προϊόντων κτλ. Το ΦΑΜ έχει σαν στόχο να δει πώς μπορούν αυτές οι δραστηριότητες να οργανωθούν πιο αποδοτικά. Παραδείγματος χάρη, αν συμφωνήσουν τα μέλη ενός ΦΑΜ ότι μία χώρα ή ένας φορέας μόναχα κάνει τον εναέριο έλεγχο για όλη την ε, ζώνη αυτό. Η άλλη χώρα αναλαμβάνει τα συστήματα μηχανογράφησης. Η άλλη ασχολείται με τα θέματα ε, προμήθειας. Είναι λοιπόν ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τους γείτονές του για να έχουμε μικρότερες οντότητες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και να είμαστε πιο αποδοτικοί. Αλλά αυτή τη στιγμή όλοι είναι στα χαρακόμματα. Κανείς δεν θέλει να δώσει ούτε ένα χιλιοστό εδάφους. Ακόμα και αν θα ήταν πιο αποτελεσματικό να έχουμε μια εναέρια διαδρομή από το α στο β στο γ για να πάει κανείς από μια χώρα σε μια άλλη. Κανείς δεν το θέλει αυτό γιατί είναι απώλεια εσόδων. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να πετύχουμε την καλύτερη λύση στη δική μας χώρα. <clears throat> Αυτό δεν είναι η σωστή αντιμετώπιση. Πρέπει να έχουμε τη σωστότερη λύση μέσα σε κάθε ΦΑΠ. Η ιδέα λοιπόν του να, συνεργαζόν, να συνεργάζονται τα κράτη μέσα στα ΦΑΠ αυτό δεν έχει προχωρήσει. Η εθνική επόπτεση είναι πάρα πολλοί συμπαθητικοί άνθρωποι, αλλά δεν έχουν καμία επιρροή και οι υπουργοί μα έχουν γραμμένους. Δεν θέλουν να τσακωθούν με τα συνδικάτα. Είπα και στα συνδικάτα των εργαζομένων. Αν δείτε πώς λειτουργεί η αεροπορική, ο αεροπορικός κλάδος. Αν κάνετε κάτι πιο αποτελεσματικό μέσα στο ΦΑΠ και κάποιοι δεν θα χρησιμοποιούνται για αυτές τις δραστηριότητες, επειδή υπάρχει αύξηση των εναρίων δραστηριοτήτων θα βρουν κάποια άλλη δουλειά. Γι' αυτό λέω στα εργατικά συνδικάτα μην αγωνίζεστε κατά της πρόοδου. Αλλά υπάρχουν οι φόβοι ότι οποιοδήποτε κινδυνεύει να χάσει τη θέση εργασία του. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε καλά παραδείγματα και γι' αυτό νομίζω ότι τα FAB όπως αυτό της Σουηδίας και της Δανίας που δημιουργήθηκε μια εταιρεία συμμετοχών και έχει λειτουργήσει καλύτερα, αυτό είναι ένα θετικό παράδειγμα. Έχουμε και άλλα παραδείγματα όπου ένα τμήμα του Υπουργείου είχε οργανωθεί σε μια χώρα με κανόνες ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία ένας κάθονται τρία άτομα μαζί που είναι ένας στρατιωτικός, ένας ιδιωτικός υπάλληλος και ένας κρατικός υπάλληλο και συνεργάζονται. Όλοι έχουν τα δικά τους κεκτημένα, τι αποδοχέ του τις διακοπέ του, Δεν θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να έχει κανεί μία δομή με την οποία να συνεργάζονται όλοι αυτοί μεταξύ του. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα αλλάξουμε όλα σήμερα. Χρειαζόμαστε όμω οδικού χάρτες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε και την ασφάλεια και να μειώσουμε την επίπτωση στο περιβάλλον. Και όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ πολιτικά. Σύμφωνα απόλυτα μαζί σου, Μπράιν οι υπουργοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά, να κάτσουν κάτω και να συζητήσουν να δουν πώς θα τα πετύχουν. Για τις τρίτες χώρες επίσης έχουμε ένα καλό παράδειγμα. Στο Φάπσι έχουμε συμπεριλάβει την Βοσνία και την Κροατία που μπήκαν με τη δική τους θέληση. Εφόσον είναι μια οργάνωση από τα κάτω, οποιοδήποτε μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον να γίνει μέλος ενός ΦΑΠ και του ρώτησα, θέλετε να προσκαλέσετε τη Σερβία. Όχι, μου είπαν αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, πολύ πολιτικά ευαίσθητο. Αλλά με τον τρόπο αυτό έχουμε μια τρύπα στα Δυτικά Βαλκάνια. Κάποιο πρέπει να έχει την πολιτική θέληση να πει εντάξει, θα του ζητήσω να γίνουν μέλο είτε του δικού μα ΦΑΜ ή κάποιου άλλου ΦΑΜ. Εναπόκειται ακόμα λοιπόν στα κράτη-μέλη, δεν είναι θέμα τη Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει απόλυτο δίκιο. Τα κράτη-μέλη επιμένουν ότι έχουν ακόμα χρόνο μέχρι το 2012 ακόμα και αν είπαν ότι θέλουν να επιταχύνουν τις διαδικασίες και παρά το γεγονός ότι ξέρουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα για να ευδοκιμήσει αυτή η διαδικασία, αλλά σας λέω και πάλι είναι θέμα των κρατών μελών τα οποία δεν έχουν δείξει ακόμα την απαραίτητη πολιτική θέληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για να είμαι ειλικρινής, <clears throat> λένε κάποιοι από τον αεροπορικό κλάδο ότι πρέπει ο επίτροπο Κάλλα να κατεβάσει ένα νέο πακέτο και να ξεπεράσει αυτέ τι αντιρρήσει των μέρων. Αλλά προσέξτε, έχουμε προχωρήσει πολύ αργά. Πρώτο πακέτο 2004, δεύτερο πακέτο 2009. Προ το παρόν Κομισιόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία που έχουμε περάσει εμεί ήδη, τα κράτη-μέλη έχουν καιρό μέχρι τι 4 Δεκεμβρίου 2012. Και αν θέλετε να έχετε ένα νέο πακέτο, που να έχει μια πιο κεντρική σχεδίαση εκ των άνω. Η Κομισιόν θα χρειαζόταν να κάνει αξιολογήσεις, να υπάρξει μια συμφωνία σε μια γενική αντιμετώπιση και δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι οι επίτροποι αυτοί θα είχαν πρόβλημα με μια τέτοια προσέγγιση, αλλά αν παρουσιάζεται ένα τρίτο πακέτο στα κράτη-μέλη, θα χρειαζόταν τουλάχιστον δύο χρόνια για να εγκριθεί και τουλάχιστον ένα χρόνο για τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ένα νέο πακέτο. Μιλάμε τώρα για πράγματα που θα γίνουν το 2015-2016, αν είναι εφικτά. Γι' αυτό λέω όχι. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να οργανώσουν τα FAB και το Κοινοβούλιο καθώς και η Κομισιόν Θα πρέπει να σπρώξουν τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό που είναι εκ της νομοθεσίας υπόχρεοι να κάνουν και γεζίνε. Σύμφωνο απόλυτα. Θα ήταν καλό σε ορισμένε περιοχές να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τους υπευθύνου των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιριών, να κάνουμε δημόσια, ε, δημόσιες εκδηλώσεις, να πείσουμε τους υπουργούς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και τη δημόσια υποστήριξη και από τον αεροπορικό κλάδο. Πρέπει, πρωτού προχωρήσουμε στο επόμενο γύρο, να κλείσουμε αυτό το γύρο. Και επομένως σας ευχαριστώ και επίσης για την Ισλανδία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τους είπα ότι αν θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σύστημά μας. Είπαν όμως ότι μέχρι στιγμής δεν είμαστε και το δικό μας σύστημα δουλεύει καλύτερα. Και έχουν ακόμα ένα σύστημα αερίου ελέγχου με τηλέφωνα και ένα σύστημα το οποίο δουλεύει σε επίπεδο από, τη μια όχθη του ωκεανού ως την άλλη. Αλλά παρόλα αυτά εγώ καταλαβαίνω και δέχομαι αυτά που είπε η Γεζίνε και άλλοι. Κάθε εθνικό κοινοβούλιο θα πρέπει να μιλήσει με τους εθνικούς υπουργού και να τους ρωτήσει τι θα προτείνετε για το θέμα αυτό. Κάποιος Ιταλός θα μπορούσε να ρωτήσει τον υπουργό του πότε θέλει να μιλήσει για το θέμα αυτό και με ποιες χώρες θέλουν να συνεργαστούν, ποιες θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους γιατί σε επίπεδο χαρτιού υπάρχουν πάρα πολλέ χώρε, στην πράξη δεν υπάρχει καμιά συνεργασία. Και στείλτε μου, αν θέλετε, ένα email και εγώ θα απαντήσω στο βαθμό που μπορώ οποιοδήποτε ερώτημά σα. Ωραία. Τώρα πάμε στον κύριο Πίτερ Γκρίφιθ, ο οποίος είναι πρόεδρος ε, του, της υπηρεσίας ελέγχου των επιδόσεων θα μιλήσει σε τεχνικό, για, τεχνικό, το τεχνικό επίπεδο και όχι για τις πολιτικές δυσκολίες. Ε, να σας πω ότι αυτή η υπηρεσία, αυτός ο οργανισμός είναι ανεξάρτητος και ελέγχει τις, ε, τις επιδόσεις και ε, καθορίζει συντελεστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που ήρθα, που μας καλέσατε. Άκουσα την συζήτηση με τον Γεώργο και προφανώς ε, μπορώ να σας απαντήσω κάποιες απορίες. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε. Όσοι δεν ξέρετε αυτό το σχέδιο, ε, το προετοιμάζουμε εδώ και ένα χρόνο περίπου. Η πρώτη έκθεση για τους στόχους ορίστηκε πέρυσι στις 27 Σεπτεμβρίου και γύρω στην ίδια ημερομηνία φέτος υποβάλαμε τα σχέδιά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή των Ενιαίων Εθέρων. Ε, βλέπετε εδώ ε, μια διαφάνεια. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να διατηρήσουμε μια, ένα οριζόντιο επίπεδο απόδοσης με στόχους ετήσιους με εξοικονόμηση 5% ε, κατ' και για να σας μιλήσουμε με, με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία Έχουμε 9,5 εκατομμύρια πτήσεις, 40.000 προσωπικό, ε, οι επιβαρύνσεις είναι 6,2 δισεκατομμύρια. Θα ξοδέψουμε γύρω στα 18,9 δισεκατομμύρια όσον αφορά την διαχείριση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να να αναθεωρήσουν κάποια σχέδιά τους ε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία υπάρχουν. Έχουμε 922 εκατομμύρια καθυστερήσεις ε, για την ε, περίοδο 2012-2004 αν δεν πετύχουμε τους στόχους μας. Επομένως ε, βλέπετε τι ακριβώς πρέπει να εξοικονομήσουμε από την παρούσα διαδικασία για FAB, διότι δεν ε, λειτουργούν τα κράτη αυτόνομα, αλλά ε, από κοινού. Ας δούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες τώρα. Όσον αφορά τους στόχους μας, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει ένα καταποκοπή κόστος όσον αφορά το το αυξανόμενο, την αυξανόμενη κυκλοφορία. Επομένως, αυτό που βλέπετε εδώ είναι το κενό ανάμεσα σε αυτό το οποίο χάσαμε στην περίοδο 12-13, ε, το, το μπλε, και το πράσινο είναι αυτό το οποίο πετυχαίνουν τα κράτη ουσιαστικά. Ε, ούτως ή άλλως για, το προηγούμενο για το, το 12-13 δεν είναι το πραγματικό στόχος, είναι ο ιδεατός στόχος που εμείς του θέτουμε. Ε, το, 2014 είναι ο πραγματικός στόχος τον οποίο επιζητάμε. Τώρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγορά μας προσπαθεί ε, να πετύχει μια καλύτερη ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια αγορά και οι στόχοι τους οποίους θέτουμε εμείς είναι απόλυτα ρεαλιστικοί. Εάν δείτε την διαφορά που υπάρχει, βλέπετε τα κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την επίδευση των στόχων. Έχουμε την Ουγγαρία, το ΦΑΜΠΑ, Δανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ισπανία, Αυστρία, ΦΑΜΠΕΚ και Ελλάδα το, για το ΦΑΜΠΕΚ πραγματικά εκπλήσωμε εάν δείτε το μέγεθος και τα κράτη στα, τα οποία συμμετέχουν. Ε, δεν πετυχαίνει το στόχο για πολύ λίγο, για πολύ λίγο 0,5% ενώ του ζητάμε 0,31%. Επομένως δεν είναι και τόσο μεγάλο το, η πολύ μεγάλη διαφορά. Στην Ελλάδα όμως μας ε, είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Βλέπετε τον γκρι. τον γκρι είναι η Ελλάδα. Mm και όμως η Ελλάδα είναι ε, πραγματικά ε, σε πολύ κέριο σημείο διότι είναι ο σύνδεσμός μας με την Μέση Ανατολή και όταν υπάρχουν καθυστερήσεις στην Ελλάδα ε, οι επιπτώσεις είναι για όλο τον ενάωριο χώρο της Ευρώπης. Και αυτό κοστίζει δυσανάλογα πολλά. Πρέπει όμως και αυτό να το διορθώσουμε. Ε, μου έκανε εντύπωση και με ευχαρίστησαν αυτά που άκουσα από, την, από τον συνάδελφο από την Τσεχία, διότι η, εάν δείτε το FAB CE, που είναι ένα πολύ σημαντικό FAB για μας, θα δείτε ότι τα κράτη τα οποία συμμετέχουν έχουν κάνει τις δικές τους ε, επενδύσεις που δεν είναι και συντονισμένες. Αν δείτε τη Σλοβενία που είναι το μικρότερο κράτος από όλα, θα δείτε ότι διπλασιάζει το κόστος κάνοντας ε, πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για μια χώρα όπου το πιο γρήγορο τζέτ την ε, περνάει σε 4 λεπτά ενώ το πιο αργό σε 8 λεπτά. Επομένως ε, πιστεύουμε ότι η συνεργασία Αυστρίας-Σλοβενίας ε, μπορεί να ανοίξει κάποιες ικανότητες έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην ε, περιοχή αυτή και με αυτό, θα, με αυτό, αυτό, το, αυτό το στοιχείο θα, θα βελτιωθεί και η ανάπτυξη στην περιοχή και το, θα λειτουργήσει καλύτερα το ΦΑΜ. Τώρα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, τη σχέση αποτελεσματικότητα και κόστους. Ε, βλέπουμε ότι το 2012 τα πράγματα ήταν καλά. Κάπω ε, δυσκολεύεται η κατάσταση το 2013 και το 2014. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, αν ε, έρθείτε σε επαφή με τους συναδέλφους σας, με τους τέλο στην στον έλεγχο ενέργεια κυκλοφορία τη χώρα σας, θα πρέπει να τους πιέσετε κάπως για να κλείσει αυτό το κενό το οποίο υπάρχει. Η Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Εστονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετωνία, Μάλτα, ε, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι χώρες, όλες αυτές οι χώρες τελικά δεν συνεισφέρουν στο σύστημα ε, επιδόσεων ε, Στην πρώτη περίοδο είχαμε πετύχει τον στόχο μας μέχρι το 2012. Το πράσινο, η πρόσινη στήλη είναι λίγο πιο ψηλή, αλλά είναι λόγοι ερμηνεία. Θα είχαμε 30 εκατομμύρια και δεν το οποίο χρησιμοποιείται. Όταν όμως αρχίζουμε το 2013 να έχουμε προβλήματα, 112 εκατομμύρια το 2013 και 157 εκατομμύρια το 2014 σε σχέση με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, τότε νομίζω ότι μπορούν τα κράτη-μέλη να ε, καλύψουν το κενό και να ε, μην υπάρχει ε, διαφορά ανάμεσα στα χρήματα τα οποία δεσμεύουμε και σε αυτά τα οποία πρέπει να επενδυθούν. Τώρα, όσον αφορά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε. Όσον αφορά τους στόχους κυρίως, είναι θέματα ασφάλειας, περιβάλλοντος και αποτελεσματικότητας, ε, σε γενικότερα ε, όσον αφορά την, ε, τους στόχους επιδόσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Βέβαια πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίω, περαιτέρω βελτίωσης ε, αν δείτε το, την ιστοσελίδα μας που είναι κομμάτι του Eurocontrol μπορείτε να, να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υιοθετήσουμε ρεαλιστικούς στόχους. Να έχουμε ένα σύστημα, δηλαδή ένα σχήμα το οποίο να είναι αποτελεσματικό μεν, αλλά να έχει και γι' αυτό να έχει ρεαλιστικούς στόχους. Εμείς προσπαθήσαμε ε, να το, το σχήμα αυτό να το υιοθετήσουμε με βάση την εμπειρία του, του, του Eurocontrol να στηρίζεται στην φιλοσοφία των ενιαίων εθέρων. Οι στόχοι αυτοί υιοθετήθηκαν το 2010 και είναι εφικτοί. Τώρα, το, τα σχέδια ε, επιδόσεων των εθνικών και μάλλον τα σχέδια των εθνικών επιδόσεων και των επιδόσεων των FAB θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνει, να γίνει περισσότερη δουλειά. Κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους και αυτό να το κάνουν και σε συνεργασία μεταξύ τους αλλά και μέχρι του χρόνου θα πρέπει ε, να έχουν γίνει οι απαραίτητες ε, διορθώσεις. Είμαστε σίγουροι ότι οι στόχοι αυτοί που έχουμε θέσει είναι εφικτοί και έχουμε κάνει 27 συστάσεις στην έκθεσή μας ε, που υποβλήθηκαν στην Κομισιό και η Κομισιό τις ενέκρινε και τις υπέβαλε στην Επιτροπή Ενιαίων Εθέρων για επικύρωση. Και είμαι βέβαιος ότι με τη βοήθειά σας μπορούμε να πετύχουμε τη διαφορά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκρίφιθ. Ας ανάψουμε πάλι τα φώτα. Υπάρχουν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής, υπάρχουν παρατηρήσεις προς τον κύριο Γκρίφιθ. Καντράουι, Φώστερ, Σαΐτ πρώτος. Σας ευχαριστώ κύριε Γκρίφιθ, για την παρουσίαση που κάνετε. Μας δώσετε κάποιες πολύ σαφείς εξηγήσεις. Κάποιες ερωτήσεις θα ήθελα να θέσω. Η σχέση με το ΣΕΖΑΡ. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην φάση αυτή για να δούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βρισκόμαστε ακόμα στην προπαρασκευαστική φάση. Deployment phase στα αγγλικά. Αυτή θα έρθει κάποια στιγμή αργότερα. Πάντως έχουν γίνει συγκεκριμένε προτάσεις. Εφόσον αφαιρόμαστε όμως το 2014 ή σε κάποια μελλοντικά χρόνια, το Σέζερ θα έχει μια επίπτωση τότε στο μέλλον και πώς θα εμπλακείτε εσείς. Ενδεχομένω ως προς αυτό να μπορούσατε να μα δώσετε κάποιε παραπάνω εξηγήσεις, κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρατηρήσει σε δύο σημεία. Στην ενδιάμεση φάση, ενώ όλα αυτά θεωρητικά προχωρούν, Φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, αν δούμε για παράδειγμα ζητήματα όπως η ακριβή αναχωρήσεων, η συμφόρηση, ότι ότι στην περίπτωση αυτή υπήρχε μια ευέλικτη χρησιμοποίηση του ενέργειου χώρου και σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία. Επομένως, και ξέρετε ότι ορισμένα κράτη-μέλη είχαν επιλύσει τα προβλήματα αυτά πρωτού καν μιλήσουμε για φάμπα. Τι γίνεται όμως με τα κράτη-μέλη αυτά, τα οποία ακόμα και στη φάση αυτή επιμένουν να μην αντιμετωπίσουν ευέλικτα τον ενέργειο χώρο ούτε για την πολιτική ούτε για την πολεμική αεροπορία. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη τώρα. Θα αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στον Ομένο Βασίλειο προχωράει το σύστημα FAB και το FAB ιρλανδια στο Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά παρόλα αυτά δεν πετυχαίνουμε κάποιους στόχους και αυτό δεν είναι αποδεκτό, κατά την άποψή μου. Και όχι μόνο επειδή, επειδή ουσιαστικά ένα 75% των επιβατών που φτάνουν στο Μένο Βασίλειο, φτάνουν από τρίτες χώρες προς το μένο Βασίλειο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ζητήματα όπως ο τουρισμός τι πρόκειται να κάνετε εσείς γι' αυτό και τι θα γίνει με τον ΝΑΤ, δηλαδή τον Εθνικό Φορέα Παροχής Υπηρεσιών στο Μένο Βασίλειο. Αναφερθήκατε σε network managers, ε, φορείς διαχείρισης των δικτύων. Δεν ακούσαμε κάτι για αυτούς μετά την ε, περίφημη περίπτωση της έκρηξης του ηφαιστείου. Σε μια ρεαλιστική βάση λοιπόν, Πίτερ, πώς πιστεύεις θα καταφέρουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά γιατί τα πράγματα δεν βαίνουν αισίω και αυτό δεν είναι καλό. Ευχαριστώ. Κύριε Γκρίφιτ, θέλετε να απαντήσετε πρώτα στι δύο αυτέ ερωτήσει και συνέχεια να δώσω και το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον θέλει και αυτή να απαντήσει. Χαίρομαι κύριε Πρόεδρε που θέσατε το πρόβλημα για το ΣΕΖΑΡ. Είναι ένα σημαντικό εγχείρημα, αλλά πρέπει να αποδώσει καρπούς και πρέπει να το κάνει αυτό στην δεύτερη περίοδο αναφοράς από το 2015 και επέκεινα γιατί αυτό το πρόγραμμα αρχίζει να γίνεται πολύ σημαντικό για μας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί σε περιοχές όπου μπορεί να κάνει τη διαφορά και αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει στο ΣΕΖΑΡ. Πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη αξιολόγηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και με τη διαδικασία IP1 που είναι τα στοιχεία πριν από το ΣΕΖΑΡ αρχίσαμε να βλέπουμε τον αντίκτυπο που θα προκύψει στις 10 Μαΐου η Κομισιόν έστειλε μια επιστολή υποστηριζοντας τις ενέργειές μας με, τους στόχους, ε, με τη στόχοθεσία για την απόδοση. Θα έπρεπε λοιπόν να μας δώσουν μια απάντηση πόσες από τις επενδύσεις αυτές είναι πράγματα που έπρεπε να γίνουν πριν εφαρμοστεί το ΣΕΖΑΡ. Ποια είναι τα στοιχεία λοιπόν από τους 80 στόχους του IP1 θα είναι στοιχεία του ΣΕΖΑΡ και ποια όχι. Δυστυχώς δεν μας έχουν απαντήσει. Ζητήσαμε λοιπόν από τα κρατη να μας απαντήσουν καλύτερα. Όταν ερχόμαστε στη δεύτερη περίοδο αναφοράς, η οποία για μας ξεκινά στις 9, στις 10 καλύτερα Νοεμβρίου, γιατί πρέπει να γίνει μια πρώιμη σχεδίαση. Θέλουμε να δούμε τι θα κάνει το ΣΕΖΑ στην περίοδο αναφοράς, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος, πώς θα υλοποιηθούν αυτά και πώς θα τα μετρήσουμε. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του ΣΕΖΑ αλλά πρέπει να γίνει σωστή καταμέτρηση των αποτελεσμάτων που μπορούν να προκύψουν από το πρόγραμμα αυτό. Αν θέλουμε να φτάσουμε τους στόχους του κεντρικού σχεδίου του Master Plan, θα πρέπει να γίνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές, γιατί ο χρόνος, όπως έλεγε και ο Δημοσθένης, μας τελειώνει. Μέχρι το 2015 θα πρέπει να έχουμε για να έχουμε το 50% που ζητάμε θα πρέπει να γίνεται μία μείωση 12,75 το χρόνο για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Για το ερώτημα της κυρίας Φώστερ, χαίρομαι που αναφέρεστε και στη στρατιωτική χρήση του εναέριου χώρου. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε σχέση με το κενό, με το έλλειμμα χωρητικότητας. Βλέπουμε και εδώ το ΦΑΜΠΕΚ παίζει ηγετικό ρόλο για να χρησιμοποιηθεί πιο ευέλικτα ο ενάριος χώρος. Όλα αυτά είναι κάπως σε εμβριακή φάση. Θα πρέπει να μεταφραστεί και στα 29 κρατη που συμμετέχουν στο σύστημα των ενιαίων εθέρων. Είμαι σίγουρο ότι πολύ περισσότερα μπορούν να γίνουν για να επιτευχθεί αυτό το θέμα. Όταν δούμε και τη διαδικασία παρακολούθηση και ελέγχου που πρέπει να εφαρμοστεί από το 2012, σίγουρα θα εξετάσουμε και κάποιου μηχανισμού για πιο ευελέκτη κρίση του ενεργείου χώρου, γιατί πρέπει να δούμε πότε οι στρατιωτικοί ε, απελευθερώνουν χρόνο, αλλά πότε ο απελευθερωμένος αυτός χώρος χρησιμοποιείται από τις πολιτικές αρχές αεροπορίας. Κάνουμε λοιπόν την αρχική εργασία του να δημιουργήσουμε το πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου και στη συνέχεια μπορούμε να ελέγξουμε λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα μετά από τον πρώτο χρόνο ε, λειτουργίας. Και για το Ηνωμένο Βασίλειο, το, το Συμβούλιο για την Αξιολόγηση της ε, απόδοσης μιλάει, έχει συνομιλητή την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι δικιά τους δουλειά να εισαγάγουν το σύστημα των ενιαίων εθέρων και έχουν προχωρήσει μέσα από μια ενδελεχή διαδικασία αναθεώρησης του κόστους και ελέγχου του κόστους. Είμαι σίγουρος ότι ο στόχος των ενιαίων εθέρων είναι κάτι που τους ενδιαφέρει. Θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους και να δούμε πώς θα μπορέσουν να επιτύχουν το στόχο αυτό. Αυτή τη στιγμή λένε ότι συζητάνε τα θέματα αυτά. Γύρω στις 20 Οκτωβρίου θα επανέλθουν σε εμά. Λοιπόν και πάλι, αν θέλετε να έχετε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί μας για να ξέρουμε τι γίνεται, σίγουρα οι συνάδελφοί μου στην Κομισιόν θα μπορούν να μας δώσουν κάποια περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Όλοι μπορούν να συζητήσουν, όλοι μπορούν να συμμετάσχουν. Εγώ χαίρομαι να έρθετε στο Ηνωμένο Βασίλειο και να συζητήσετε και αν θέλετε υποστήριξη από μένα θα την έχετε. Για τον ε, διαχειριστή δικτύου. Έχει ανασκουμπώσει τα μανίκια του φέτος και πολλή δουλειά. Δεν ήταν το θέμα αυτό που αναφέρατε μονάχα με το ηφαίστειο στην Ισλανδία, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει τις γενικές καθυστερήσεις, κυρίως στην Αυστρία και στην Κύπρο, όπου υπήρξε μεγάλη πίεση ενάρειας κυκλοφορία, έχει μειωθεί τελικά αυτή η καθυστέρηση. Και αν συνεχίσουμε την πορεία αυτή βελτίωση της διαχείρισης στις δύο αυτέ χώρες, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο του 0,5. Αυτά λέει η αξιολόγηση. Επομένως, ο διαχειριστής δικτύου αρχίζει να είναι αξιόπιστος, αρχίζει να έχει αποτέλεσμα. Χρειάζεται όμως περισσότερο χρόνο για να μπορέσει να διατυπώσει σχέδια επί τη βάση του συνόλου δικτύου. Ελπίζουμε λοιπόν το Μάρτιο του 2012 θα μας πει ο διαχειριστής δικτύου ποια είναι η στρατηγική του ώστε να μπορούμε μέχρι, τις, μέχρι τον Ιούνιο του 2012 να έχουμε την αναθεώρηση και τη στρατηγική μας και αν χρειάζεται να προτείνουμε τροποποίηση. Αλλά είναι σημαντικός ο ρόλος του διαχειριστή δικτύου και θα πρέπει να δώσει καρπούς η προσπάθειά του. Εντάξει λέει ο πρόεδρος Σίμψον. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον κύριο Γκρίφιτς και τον Γκέορκ για τη σημερινή τους παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ εμπλουτιστικά αυτά για τη συζήτηση και μας κατέδειξε που πρέπει να προχωρήσουμε ως πολιτικοί για να καλύψουμε τις πολιτικές ανάγκες στο θέμα αυτό. Μπορώ να δω λοιπόν ο Τζάκι να διατυπώνει ένα γράμμα στην Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ουσιαστικά πρέπει να ασκήσουμε πίεση στι εθνικέ μα αρχέ και στου εθνικού μα υπουργού για να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουν κάτι για αυτό το FAB το οποίο όλοι το υπέγραψαν. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε εν καιρό. Ευχαριστώ. I'm now just going to ask shortly because... Τώρα. Αυτά τα λουλούδια είναι για τον Τζέραλτ. Αλλά η Σίλβια ήθελε να τα δώσει αυτά τα λουλούδια, γι' αυτό θα ζητήσω από την Αντιπρόεδρο να μας να δώσει τα λουλούδια στον Τζέραλτ. Καλύτερα τα κάνει μια ωραία γυναίκα όταν δίνει λουλούδια παρά ένας άσχημος άντρας, λέω, ο πρόεδρος. Εντάξει. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα τη ημέρας διάταξη που είναι η ιδία μου έκθεση σε σχέση με το Μνημόνιο συνεργασία με την ΙΚΑΟ, τη Διεθνή δηλαδή Οργάνωση πολιτική Αεροπορίας, για να σας δώσω το γενικό πλαίσιο. <clears throat> να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν κάπου 190 κράτη-μέλη στον ΙΚΑΟ και συνεργάζονται, υποτίθεται ότι συνεργάζονται τουλάχιστον, στον τομέα της ασφάλειας, της εναερίες μεταφορές, της προστασίας των αεροπορικών ε, ε, συγκοινωνιών, της καλύτερης διαχείρισής του κτλ. Τα πρότυπα της ΙΚΑΟ ε, έχουν ενσωματωθεί στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματος χάρη τα, τα πρότυπα για το περιβάλλον και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στο να μπορέσει να συμβάλλει στην διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής στον ΙΚΑΟ. Και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βοηθά και την ανταγωνιστικότητα της δικής της πολιτικής αεροπορίας. Το Μνημόνιο συνεργασία έχει σαν στόχο να κάνει επίσημη τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΙΚΑΟΥ και ιδίω θέλει να εξασφαλίσει καλύτερη αναμόνιση προτύπων και καλύτερο συντονισμό για τι αντίστοιχε δραστηριότητε. Ο στόχο μα επίση είναι να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο του περιορισμένου πόρου μας και να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Η συνεργασία περιλαμβάνει συμφωνίε για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει εμπειρογνωμοσύνη και πόρου στο ΙΚΑΟ και παρατηρητέ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμμετέχουν σε αποστολέ ελέγχου του ΙΚΑΟ στα κάτι μελη Επίση, σύμφωνα με του εφαρμοστέου κανόνε, τα συμβαλώμενα μέρη θα ανταλλάσσουν ηλεκτρονικέ πληροφορίε, δεδομένα και επίσημε δημοσιεύσει και θα παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε βάσει δεδομένων. Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου εγκρίνει το μνημόνιο αυτό και θεσπίζει μια κοινή επιτροπή που θα είναι το αρμόδιο σώμα για την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας. Συνεργασίας είπα και καθορίζει τις συγκεκριμένες διαδικαστικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή του Συμβουλίου της Κομισιόν και των 100 μελών μας στα πλαίσια της Επιτροπής. Επιπλέον, υπάρχουν ρυθμίσει σε σχέση με συγκεκριμένου τομεί συνεργασία που θα προσαρτηθούν στο μνημόνιο και θα αποτελέσουν αναπόδραστο και αναπόσπαστο τμήμα του. Για να βρούμε ποιοι είναι οι τομεί όπου υπάρχει έλλειψη ασφάλεια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι αεροπορικέ εταιρείε και πολύ σημαντικό στοιχείο τη κοινή μα δραστηριότητα. Γι' αυτό το Συμβούλιο έχει επιφορτήσει την Κομισιόν να θεσπίσει διατάξει που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των αερογραμμών. Αυτέ οι ρήτρε θα πρέπει να δημιουργηθούν με κοινή δράση και συντονισμό μεταξύ των συμβαλωμένων μερών. Η προσέγγιση βασίζεται στην κοινή δέσμευση να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο σε παγκόσμιο επίπεδο αεροπορική ασφάλεια και ένα παγκόσμιο εναρμονισμό των ε, κοινών πρακτικών και των προτύπων ασφάλεια. Στι 16 Ιουνίου το Συμβούλιο ενέκρινε αυτό το παράτημα για την ασφάλεια των αεροπορικών συγκοινωνιών, το οποίο ενεκρίθη επίσημα από μια μεικτή επιτροπή. άλλη τομή συνεργασία, η ασφάλεια στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Η διαχείριση της κυκλοφορίας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω παρατημάτων. Επειδή βάσει μιας πρότασης της Κομισιόν, το, το Συμβούλιο θα καθορίσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στη Μικτή Επιτροπή. Τα παρατήματα αυτά δυστυχώς δεν θα υπόκεινται στη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου γιατί το άρθρο 218 παράγραφος 9 δεν προβλέπει οποιαδήποτε συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής με τον ΙΚΑΟ. Αλλά ο εισηγητής σας, ο υποφαινόμενος, θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμβάλλει σε μια πιο στεναρή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στον ΙΚΑΟ και σε ένα πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας και προτείνει ως εκ τούτου ότι η Επιτροπή Μεταφορών θα πρέπει να δώσει την έγκρισή της σε σχέση με τη σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας. Υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να δίνει την σύμφωνη γνώμη του στην περίπτωση αυτού του Μνημονίου με μία και μόνο ψηφοφορία δεν μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες ή θα πούμε ναι ή θα πούμε ου. Αυτά είναι η έκθεσή μου λοιπόν. Ο κύριος Γκρός θέλει πει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά θα υποστηρίξουμε την πρότασή σας και θα υποστηρίξουμε με ναι την πρότασή σας. Έχω μόνο μερικά ερωτήματα σε σχέση με τη, συμφωνία, τη λεγόμενη συμφωνία του Σικάγο που εμπλέκεται σε πολλούς τομείς όπως παραδείγματος το θέμα της συγχωρήπανσης από τα αεροπλάνα. Εγώ δεν έχω <clears throat> πρόβλημα ως κοινοβούλιο να συμμετάσχω σε αυτό το έργο, αλλά θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν και εκ των προτέρων μπορούσαμε να έχουμε πληροφορίες μέσω της Κομισιόν για τα θέματα αυτά, γιατί υπάρχουν και πολλά ζητήματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο συζήτησης για μας, όπως είναι η ενάρια ασφάλεια και το περιβάλλον και τα οποία φυσικά τη χάνουν επεξεργασία συγχρόνως και σε διεθνές επίπεδο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για το Κοινοβούλιο να μπορούμε να έχουμε γνώσεις για τα διαμοιβόμενα στον διεθνή αυτή, αυτό φορέα του ΙΚΑΟ. Θυμάμαι ότι έχουμε μιλήσει πολλές φορές για πολλά θέματα ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής όπου δεν είχε υπάρξει μια τεράστια εμπιστοσύνη και από, από τις δύο πλευρές εδώ νομίζω ότι έχουμε μεγάλε δυνατότητε να πληροφορηθούμε για επερχόμενες συμφωνίες στον τεχνικό δρόμο, είτε με άμεση πληροφόρηση, είτε μέσω τη Κομισιόν. Αυτή θα ήταν η πρώτη μου πρόταση και το ερώτημα του αν αυτό είναι εφικτό βέβαια είναι το ερώτημά μου. Και το δεύτερο, και εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε φορεί οι οποίε ασχολούνται με τα θέματα τη ενάρεια ασφάλεια, Πώς εμπλέκονται εδώ στη δομή αυτή που αναφέρεται ή το έργο τους είναι τελείως παράλληλο με αυτό του που καλύπτεται από το μνημόνιο συνεργασίας και προκύπτει πρόσθετο κόστος και άχρηστη δαπάνη ανθρώπινης ενέργειας ή είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν μια καλύτερη συνεργασία. Και πάλι μια πρόταση και μια ερώτηση είναι αυτό το οποίο σας λέω. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς, το Κοινοβούλιο καλείται να δώσει την σύμφωνη γνώμη του στο, στην ολοκλήρωση του Μνημονίου Συμφωνίας. Είναι ένας συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Διεθνούς Οργάνωσης ε, Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι πολύ σημαντικό κείμενο. Ο εισηγητής είπε τα πάντα. Απλώς ε, θα ήθελα να πω ότι και η ομάδα μας, οι φιλελεύθεροι, συμφωνούν απόλυτα και να προσθέσω απλώς τρεις σκέψεις μου. Καταρχάς, οι περισσότερες, τα περισσότερα από τα πρότυπα του, της ΔΟΠΑ, του ΙΚΑΟ δηλαδή, ήδη έχουν συμπεριληφθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία νομοθεσία. Ε, και θα πρέπει τα και τα υπόλοιπα να τα εντάξουμε στην νομοθεσία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στην, στον καθορισμό και στο σχεδιασμό των πολιτικών τη Διεθνού Οργάνωση πολιτική Αεροπορία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, να το παραμελήσουμε. Τώρα θα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι άλλο το οποίο ε, ε, αρέσει πολύ στην, στην Άλντε είναι η απλούστευση των διαδικασιών με ένα το πλεονέκτημα να έχουμε ένα και μόνο εργαλείο το οποίο θα καθορίζει τον ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμών έναντι της ΔΟΠΑ. Ε, κάτι, ένας τρίτος λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι είναι ε, πολύ θετική η σύναψη αυτής της συμφωνίας είναι ε, ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την διαφάνεια και την, όσον αφορά τις διαδικασίες, όσον αφορά και την χρηματοδότηση, τον προϋπολογισμό. Παραδείγματο χάρη, την μεταφορά των πόρων από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση στην γραμματεία της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας. Η κυρία Φώστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εξηγήσει. Σε γενικές, γενικές γραμμές υποστηρίζω αυτά τα οποία είπατε. Πιστεύω ότι η ΔΟΠΑ, η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, είναι ένας ισχυρός οργανισμός. Είναι μια επισημοποίηση, αν θέλετε, αυτού του, ε, του, του status quo, αυτό του οποίου ήδη συμβαίνει εδώ και καιρό καλό θα είναι να υπάρχει εναρμόνιση και επιβολή ενιαίων προτύπων στο συγκεκριμένο τομέα. Ταυτόχρονα όμως ε, είναι απόλυτα κατανοητό και το κοινοβούλιο δεν είναι υποχρεωτικό να παρεμβαίνει, διότι 190 χώρες μετά θα πρέπει να πούνε τις απόψεις τους, 190 κοινοβούλια. Τέλος πάντων, θα πρέπει γενικότερα να προωθήσουμε τέτοιου είδους συμφωνίες. Όπως είπε και η Κομισιό, τα πράγματα έχουν προχωρήσει, είναι, έχει επισημοποιηθεί η σχέση πλέον και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ θετικό, διότι μιλάμε για μια διεθνή, ένα διεθνή κλάδο πλέον. Uh, Κύριε Τικά, σας ευχαριστώ. Μία ερώτηση θέλω να θέσω το πρωτόκολλο αυτό, το μνημόνιο αυτό συνεργασίας, πρόκειται να επιφέρει κάποιες θετικές αλλαγές όσον αφορά το σύστημα πολιτικής αεροπορίας και ποια θα είναι η διασύνδεσή του με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ε, εκπομπής. Πρωτό απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα υπάρχει και ένα επιπλέον παράρτημα το οποίο θα έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Η δικιά μου ανησυχία είναι ότι όταν προσαρτηθεί αυτό το παράρτημα εμείς δεν θα μπορέσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πειράσουμε καθόλου τα πράγματα. Δεν θα έχουμε λόγο γι' αυτό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μαντέψουμε μια κάποια λύση για το ETS. Αν εσείς έχετε κάποια ιδέα, σας παρακαλώ πολύ να μου το πείτε κύριε Σίμπο. Να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί δεν σε έδωσα το λόγο όταν ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τα ΦΑΜΠ. Έπρεπε να σας δώσω τότε το λόγο. Αν θέλετε να μιλήσετε για τα ΦΑΜΠ, παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους όσοι συνέβαλαν στην ε, συζήτηση αυτή. Το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτό που και ο συγγητής πάρα πολύ καλά, ποια είναι η βασική διαδικασία πίσω από αυτό το μνημόνιο συνεργασία. Είναι ένα μνημόνιο το οποίο ενδυναμώνει και διευκολύνει τη συνεργασία μας με έναν πολύ σημαντικό υποοργανισμό των ΗΠΑ Εθνών, δηλαδή τον ΙΚΑΟ, τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν θέλω να αποφύγω την τελευταία ερώτηση που έγινε που έχει να κάνει με το ETS. Σαφώς γνωρίζετε ότι εδώ πέρα έχουμε κάποια προβλήματα. Δεν καταφέρνουμε να πείσουμε διμερός και πολυμερός τους εταίρους μας ανά τον κόσμο για την χρησιμότητα, την καλή βάση της νομοθεσίας αυτής. Τίθεται όμως ένα γενικότερο πρόβλημα. Στα πλαίσια του ETS δεν είναι πρώτη φορά που συναντούμε προβλήματα στη συνεργασία που έχουμε με τον ICAO σε σχέση με την υφιστάμενη τη νέα κοινοτική νομοθεσία και την συνεργασία έπειτα που έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΙΚΑΟ. Πριν από δέκα χρόνια θα θυμάστε ότι ε, είχαμε ένα άλλο πρόβλημα με κάποια αεροσκάφη. Βρισκόμαστε αστικά στην ίδια κατάσταση με αυτή που αντιμετωπίσουμε τώρα με το ETS. αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος σε πολυμερές και σε διμερές επίπεδο συζητεί το, τμήμα αυτό λοιπόν της κοινοτικής νομοθεσίας υπέρ του περιβάλλοντος και στο τέλος αναγκαστήκαμε να αποδεχθούμε κάποιες σημαντικές αλλαγές και τροποποίησεις προκειμένου να σταματήσει αυτή η διεθνής διένεξη που είχε προκύψει. Ποια είναι τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε από όλη αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέψει να καταφέρουμε να επηρεάσουμε περισσότερο την εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στον ΙΚΑΟ όσον αφορά τις συμφωνίες σε πολυμερές επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό να συνάδει η όλη αυτή η εργασία με την υφιστάμενη κοινοτική και την προτινόμενη κοινοτική νομοθεσία και ένας από τους στόχους αυτού του μνημονίου συνεργασίας είναι να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχουμε περισσότερο και να διαμορφώνουμε την πολιτική του ΙΚΑΟ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα ιδιαίτερος τώρα να αναφερθώ σε κάποιους εταίρους μας παγκοσμίως οι οποίοι Ήδη παρέχουν ε, προσωπικό, ανθρώπινου πόρου, ε, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στον ΙΚΑΟ προκειμένου να υποστηρίξουν τη την εργασία τη γραμματεία του ΙΚΑΟ. Καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη αυτή τη στιγμή δεν επεμβαίνει με τρόπο πάρα πολύ ορατό, μολονότι βέβαια υπάρχει μια κοινοτική νομοθεσία η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μέσω λοιπόν αυτού του μνημονίου συνεργασίας θέλουμε να διευθετήσουμε το πρόβλημα αυτό της ορατής συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα θέλαμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα αποθαρρύνει την επικάλυψη εργασιών. Ξέρετε ότι ο ΙΚΑΟ έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο επιτήρηση όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως κάνουμε ακριβώς την ίδια για το, την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε να συγκεράσουμε κάπως τα δύο αυτά συστήματα προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν επικαλύψεις. Και θα ήταν καλό να υπήρχε και μια ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα πορίσματα της εποπτείας αυτής. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη της Επιτροπής σας κύριε Πρόεδρε και προφανώς επιβεβαιώνω την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα φροντίσουμε να κρατάμε τη δική σας Επιτροπή ενήμερη για τις ενεξελίξει εργασίες καθώς επίσης και για την υλοποίηση αυτού του μνημονίου συνεργασίας και η ενημέρωση αυτή θα γίνεται πριν και μετά τις συνεδριάσεις της κοινή Επιτροπής. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχετε μια πλήρη εικόνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Προθεσμοί για τροπολογίε 21 Οκτωβρίου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τροπολογίε στην ίδια τη συμφωνία. Δεν ξέρω που θα τις βάζαμε λοιπόν στις τροπολογίες. Πάση περιπτώσει 22 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε και, και τον Ιανουάριο του 2012 στην Ολομέλη. Ευχαριστώ λοιπόν για τη διεκπαιρέωση αυτού του θέματος. Το επόμενο είναι η Λευκή Βίβλος για το μέλλον των μεταφορών. Φυσικά είναι ο κύριο Γκρό, ο αρμόδιος και ο εισηγητής και έχετε το λόγο κύριε Γκρός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για, για το έντονο και μερικές φορές υπερβολικά έντονο ενδιαφέρον που δείξανε για αυτό το θέμα με 413 τροπολογίες. Ίσως δεν σπάσαμε το σημερινό πρωινό ρεκόρ, αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό το ρεκόρ. Εγώ προσωπικά Έχω καταθέσει πολύ λίγες τροπολογίες γιατί ήθελα φυσικά να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα βλέποντας τις τροπολογίες των συναδέλφων να καταθέσουμε να καταθέσω κάποιες τροπολογίες συμβασμού θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταθέσει ένα συνεκτικό μήνυμα και όχι ένα υπερβολικά μακροσκελή κατάλογο μικρών διεκδικήσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσω να το επιτύχω αυτό και φυσικά θα το κάνω αυτό χάρη ελπίζω στην ε, στενή συνεργασία με τους ε, σκιώδες εισηγητές από τα άλλα πολιτικά κόμματα αλλά και με τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν καταθέσει πολλαπλές τροπολογίες. Έχει αρχίσει αυτή η προπαρασκευαστική εργασία εξάλλου ήδη. Και πράγματι πολλές ε, τροπολογίες έχουν σημασιολογικό μονάχα σημασιολογικά απλώς χαρακτήρα, θέλουν απλώς να διευκρινίσουν κάτι καλύτερα το οποίο περιέχεται στο έγγραφο. Σε σχέση με τη στοχοθεσία, η δική μου πρόθεση και πρόταση θα ήταν να προσπαθήσουμε στην έκθεσή μας να εστιάσουμε σε μια πιο σύντομη χρονική περίοδο, στην περίοδο 2011-2020, κάτι θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και επίσης να έχουμε σαφή θέση στόχων, ακόμα και σε αριθμητικούς όρους, σε ποσοστά, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν σε λευκές βίβλους έχουμε αποδηθεί σε θεωρητικά και ακαδημαϊκά ε, πονήματα τα οποία μαζεύουν, στο, μαζεύουν σκόνη στις βιβλιοθήκες, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και απτοί. Είναι σημαντικό το θέμα της ενέργειας το οποίο μας ενδιαφέρει. Εγώ δεν έχω αναφερθεί ιδιαίτερα στο σημείο αυτό βέβαια, αλλά <clears throat> είπα και κάποιο σημείο το οποίο θα μπορούσαμε ίσως να το διευκρινίσουμε καλύτερα με τους συναδέλφους. Εγώ θεωρώ ότι ιδιαίτερα στον αστικό χώρο η προσπάθειά μας θα ήταν να μην ε, ε, δηλητηριαστούμε από τη ρήπανση των πόλεων, να μπορούμε να αναπνέουμε τον αέρα. Επομένως το θέμα της κινητικότητος ε, να προωθηθεί περισσότερο. Εγώ βέβαια δεν θεωρώ ότι μόνο η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας θα λύσει το πρόβλημα, γιατί πρέπει να δούμε και από πού προέρχεται ο ηλεκτρισμός και πώς παράγεται. Αλλά αυτός ο τομέας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο να συζητηθεί πλήρως σε τεχνικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλές ε, τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στις ε, ευρύτερες περιφέρειες και τη διαμεθοριακή συνεργασία. Δεν πρέπει να σταθούμε μοναχα λοιπόν στο θέμα των συγκοινωνιών και των μεταφορών στον κεντρικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ευρύτερο χώρο ο οποίος περιλαμβάνει και τις περιφερειακές χώρες και πόλεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και θα προσπαθήσω να το εκφράσω με μια συμβαστική τροπολογία. Ευαίσθητα θέματα όπως είναι ο χρόνος οδήγησης και ο χρόνος ε, ανάπαυσης για τους οδηγούς παραδείγματος χάρη. Έχουμε ήδη μια εμπειρία από τα θέματα αυτά που ίσως ήταν οδυνηρή. Εγώ θεωρώ ότι η εφαρμογή σε ορισμένες χώρες έχει λειτουργήσει με λανθασμένο τρόπο. Έχουμε προσπαθήσει να θεσπίσουμε μία ενιαία ρύθμιση από 27 διαφορετικές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη αλλάζουν τις 27 αρχικές τους ρυθμίσεις. Ίσως χρειάζεται να έχουμε μία καλύτερη ενασχόληση με το θέμα αυτό και με κάποιες από τις τροπολογίες μας είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε στο Συμβούλιο ότι οι προθεσμίες εφαρμογής πρέπει να τηρούνται. Και επίσης σκέφτομαι και τις επιχειρήσεις οι οποίες ε, ασκούν τις μεταφορές και οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η ευελιξία γίνεται μέσα στα πλαίσια του νόμου και των κανονισμών και οι υπηρεσίες ε, επιμελητίας οι οποίες παράγονται, παρέχονται παρέχονται μέσα στα πλαίσια αυτά των οδηγιών. Για το καμποτάζ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μας ενδιαφέρει όμως παράλληλα η, το άνοιγμα των αγορών να μην γίνεται με οποιοδήποτε κοινωνικό τίμημα. Δεν μπορούμε από τη μία πλευρά να ζητάμε να υπάρχει σωστή κατάρτιση και καλές αποδοχές και την άλλη μέρα να αφήνουμε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία, καμία σχέση με το επάγγελμα και έρχονται με μισθούς dumping και χωρίς την απαραίτητη κατάρτιση να μπαίνουν στην αγορά. Αυτό θα δώσει ένα πολύ κακό ε, αποτέλεσμα για τις αγορές. Σε ό,τι αφορά τη διατροπικότητα και τον στόχο αυτό που αποτελεί για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ήδη από το 2000 μας είχε απασχολήσει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές αρχές μας και να προσπαθήσουμε, όπως είπαμε, μέσα στο στόχο αυτό για το 2010 <clears throat> να τονίσουμε ότι πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός ευρωπαϊκού δικτύου. Ξέρουμε ότι έχουμε λιγότερα σχέδια και καλύτερη υποστήριξη στα σχέδια αυτά, τα πράγματα είναι καλύτερα. Το επίπεδο της, ε, της υποστήριξης, αν είναι 30% ή κάτι άλλο μπορούμε το συζητήσουμε, αλλά λιγότερα σχέδια είναι καλύτερα από ένα ατελείωτο κατάλογο διεκδικήσεων για μεμονωμένα σχέδια και υποδομές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή την αρχή την έχουμε εγκαθιδρύσει ήδη στο παρελθόν το 2010 και νομίζω ότι χωρίς να σοκάρουμε άλλες επιτροπές όπως είναι η Περιφερειακή Επιτροπή, η οποία τώρα επανέρχεται με ορισμένες τροπολογίες που αφορά την χρήση των περιφερειακών ταμείων για την πρόθεση κινητικότητας. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά επίσης τις <clears throat> λειτουργίες των λιμένων και τις ε, υπηρεσίες των ε, λιμένων, εδώ δεν πρόκειται για ένα άκρατο άνοιγμα των ε, υπηρεσιών των λιμένων, Αυτό το θέμα είχε ήδη ε, συζητηθεί στο παρελθόν και η Επιτροπή μας είχε προετοιμάσει και μια γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να είναι και η βάση για μια νέα ε, επεξεργασία ώστε να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια άλλη αρνητική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ότι πρέπει αυτό το άνοιγμα της αγοράς των λιμένων να εξασφαλίζει και την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι για μένα δεδομένο. Ελπίζω λοιπόν ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα από διαβουλεύσεις και συζητήσεις και από συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα μεγάλο αριθμό συμβιβαστικών τροπολογιών ώστε να μειωθεί ο αριθμό των ε, τροπολογιών που θα πρέπει να επεξεργαστούμε χωρίς να παραμεληθεί το στοιχειώδες και το βασικό τους ε, περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ισηγητά και έχουμε έναν μεγάλο κατάλογο μιλητών όλκα αναλόγα για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι και άλλοι συνάδελφοι θα αναφερθούν στις τροπολογίες, επομένως δεν θα ήθελα να επισέλθω σε πάρα πολλές λεπτομέρειε. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών, μολονότι το όλο εγχείρημα είναι πολύπλοκο. Και για αυτό το λόγο λοιπόν πιστεύω ότι έχουν τεθεί κάποιοι φιλόδοξοι στόχοι στη Λευκή Βίβλο και τους στόχους αυτούς έχει συμπληρώσει ο κύριος Γκρός, ο συγητής μας. Θα πρέπει να βασιζόμαστε σε μια πολύ καλή γνώση της κατάστασης και να έχουμε ένα συγκεκριμένο όραμα για το κοντινό και απότερο μέλλον. Ζητήματα όπως η συντροπικότητα, η διασφάλιση της ασφάλειας, οι κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών είναι ορισμένα στοιχεία τα οποία έλαβε υπόψη ω σκιώδης για την ηγήτρια για την προετοιμασία των τροπολογιών. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατό να, δυνατό να κάνει μία ανάλυση τη ποιότητα και του εύρου των δικτύων μεταφορών στα κράτη-μέλη. Με τον απολογισμό αυτό θα καταφέρουμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την ασφάλεια. Για τις οδικές μεταφορές ξέρετε ότι ένα 70% των ατυχημάτων γίνονται ακριβώς στους δρόμους είτε στην Ήπεθρο είτε στις πόλεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό της ασφάλειας. Θα ήθελα επίσης ο εισηγητής να διατηρήσει ένα ενδεικτικό όριο, μια οριακή τιμή 300 χιλιόμετρων για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές, όπως ακριβώς λέγεται και στη Λευκή Βίβλο. Σαφώς θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τις βιώσιμες μεταφορές σε πιο σύντομες αποστάσεις. Ωστόσο, όσον αφορά τις μεγάλες αποστάσεις, θα πρέπει να έχουμε μια πιο συστημική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δική μου πολιτική ομάδα στις τροπολογίες που κατέβαλε επικεντρώθηκε κυρίως στην βιώσιμη αγορά εργασίας, στα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μία μελέτη αντικτύπου όσον αφορά την εξέλιξη της αγοράς εργασίας στον τομέα των μεταφορών, καθώς επίσης και μία ανάλυση όσον αφορά την ποιότητα των προτινόμενων θέσεων εργασίας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε μέχρι το 2020 τι προβλέπεται όσον αφορά την κατάρτιση, την εκπαίδευση των εργαζομένων. Πολλοί συνάδελφοι και εγώ έχουμε υπογραμμίσει στις τροπολογίες μας τις ε, διάφορες μορφές των αστικών μετακινήσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα μαζικά μέσα μεταφοράς, θα πρέπει να είναι προσβάσιμα αυτά στους χρήστες όσον αφορά το ωράριο για παράδειγμα των μεταφορών αυτών, αλλά όσον αφορά ακόμα και την τιμή τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε επίσης και τα μέσα αυτά μεταφοράς, τα οποία είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Αν θέλουμε να θέσουμε φιλόδοξους στόχους, αν θέλουμε πραγματικά να προτείνουμε προς το Συμβούλιο μία στεναρή στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να θέσουμε στόχους που θα μας επιτρέψουμε να σημειώσουμε πρόοδο και που θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμφανιστεί τελικά με μια μεγάλη πλειοψηφία στον φάκελο αυτό. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, ας μην ζητήσουμε μια εναρμόνιση των μισθών στον τομέα των μεταφορών, ας μην επιμείνουμε ιδιαίτερα στις λιμενικές υπηρεσίες, ας μην δημιουργήσουμε εμπόδια. Πρόεδρος, οι ε, διερμηνείς ζήτησαν να μιλάτε λίγο πιο αργά. Αναφερθήκαμε επίση και στην ε, οδηγία για το χρόνο εργασία, πολύ σημαντική για την ασφάλεια των οδικών μεταφορών. Πέρα από όλα αυτά όμω τα επιμέρου τμήματα πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην ε, επιτυχή εφαρμογή τη οδηγία αυτή. Να αναφερθώ και στι τροπολογίε ε, του εισηγητή. Στην έκθεσή σα έχετε αλλάξει την ημερομηνία για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Αναφέρεσαι στο 2013 αντί για το 2015. Αναφέρεστε επίσης και στον χάρτη των δικαιωμάτων ε, των επιβατών. Τέλη 2012 λέτε αντί το 2013. Γιατί το κάνετε αυτό, είστε ξαφνικά πιο αισιόδοξο σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω σε μια θετική συνεργασία στο μέλλον. Ο κύριος Γκρός είναι αιώνια αισιόδοξος. Μάισνερ, κυρία Μάισνερ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, μου είχαν ε, πει στη Γερμανία σε κάποια συζήτηση ότι μια λευκή βίβλος είναι ένα ευχολόγιο ουσιαστικά και δεν γνωρίζει κανείς ποια είναι και αυτή η χρησιμότητα μιας λευκής βίβλου. Δεν είναι ένα νομοθέτημα, αλλά είναι με ένα έναυσμα τουλάχιστον να μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερα προς ποια κατεύθυνση μπορούμε να πάμε το, στο μέλλον και μια λευκή βίβλος καλύπτει πολλούς τομείς, ακόμα και πολλούς τομείς εκτός των μεταφορών. Έκανε πολλές... Ε, ε <clears throat> είπε ο Ματιώτη ότι έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες στην έκθεσή του, 413. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές τροπολογίες, καμιά σαρανταριά, παρά το γεγονό ότι δεν είμαστε τόσοι πολλοί, είμαστε ένα τέσσερα άτομα εδώ. Θεωρούμε ότι είναι πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν στις μεταφορές. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία πολλές από τις τροπολογίες μας αφορούν τα θέματα της χρηματοδότησης, γιατί η χρηματοδότηση των οδικών, των μεταφορικών υποδομών και θεωρούμε ότι παίζει μεγάλο ρόλο η υποδομή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς θα προχωρήσει και η συνεργασία με τον εισηγητή για να μπορέσουμε να σφυριλατήσουμε τροπολογίες ε, συμβιβαστικού χαρακτήρα. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για τα ποσοστά χρηματοδότηση περισσότερα για τους, ε, ε για τους ιδεοδρόμους ή για τις θαλάσσιες μεταφορές, ακόμα και για την κυκλοφορία με ποδήλατο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν να τα σκεφτούμε καλύτερα σε επίπεδα ποσοστών χρηματοδότησης. Δεν έχουμε απεριόριστα χρήματα, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε όσο μπορούν περισσότερα κονδύλια, αλλά πρέπει να τα κατανείμουμε σε κάποια στιγμή. Αυτό λοιπόν για τα χρηματοδοτικά και για τα TNT, Αναφέρθηκε πάρα πολύ η πολυτροπικότητα και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ καλό, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες μεταφορών. Αναφέρθηκε επίσης και η δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω πολυτροπικών πλατφορμών, αλλά θα πρέπει να δούμε καταρχήν τι γίνεται με τους κύριους διαδρόμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντυπωσιάστηκα τώρα και για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περισσότερες τροπολογίες για την ε, μείωση της χρήσης ορισμένων μεταφορικών φορέων που συνδέονται με τις εκπομπές διοξιδίων του άνθρακος. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ρεαλιστικές προτάσεις για να εξασφαλίσουμε τη μείωση των πιο ρηπαντικών τομέων μεταφοράς. Και γενικά εμείς από την πλευρά των φιλελευθέρων έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ στα θέματα των λιμένων. Πολλοί από εμάς ζούμε σε παράκτιες περιοχές και επομένως νιώθουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Ε, Ματιέ, μας εξήγησες τι θέλεις να κάνεις με τις λιμενικές υπηρεσίες. Είναι πάρα πολλοί από εμά που θέλαμε να αποφύγουμε ένα νέο πακέτο με τη λογική ότι ό,τι έρχεται πολλές φορές είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Αλλά πιστεύουμε ότι με τις συμβαστικές τροπολογίες μπορούμε να έχουμε ένα θετικό δρόμο. Επίσης, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα των ε, ατόμων με αναπηρίες στις αεροπορικές ε, ε, συγκοινωνίες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μα έχει ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμεί κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε αυτέ τι συγκοινωνίε. Επίση, για τι ημερομηνίε τα πράγματα είναι φιλόδοξα γιατί ο Ματιού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φιλόδοξος. Θέλουμε να προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα από ό,τι μας προτείνει η Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα να δω πώ θα μπορέσουμε να συμφωνούμε και φυσικά πρέπει να μείνουμε πάντα στα πλαίσια του ρεαλισμού. Και χαίρομαι για τη δυνατότητα να έχουμε περαιτέρω διαβουλεύσει με τον εισηγητή. Bradburn από τους συντηρητικούς. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι συνάδελφοι ίσως θα θυμούνται ότι όταν ε, ξεκινήσει την συζήτηση αυτή ε, είχα πει ότι το κείμενο αυτό είναι εν μέρη καλό. Έχει ορισμένα καλά κομμάτια και ορισμένα όχι πολύ σωστά είπαμε, ανεφέρθηκε μάλλον, ότι δεν είναι νομοθετικό κείμενο αυτό και εγώ ευγνωμονώ και όλες το θεωρεί δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, στις τροπολογίες που έχω υποβάλει, αυτό το οποίο προσπαθώ να πετύχω είναι να τροποποιήσω ή να διαγράψω κάποια, κάποιες από τις κακές αν θέλετε προτάσεις της ε, Κομισιόν. Και ο κύριος Γκράσ στις αρχικές του παρατηρήσεις αναφέρθηκε στο σημείο αυτό και είναι απόλυτα λογικό. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια λευκή βίβλος η οποία να ασχολείται με πρακτικούς και εφικτούς στόχους και όχι ευσεβείς πόθους. Και συμφωνώ απόλυτα ματιά με αυτό το οποίο είπες ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ε, ίσως όχι τόσο μακροπρόθεσμο το, το, σχέδιο αυτό, διότι όσο πιο ε, μακριά κοιτάμε, τόσο λιγότερο εφικτή είναι η στόχη μας. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ε, μεσοπρόθεσμους, αν θέλετε, και εφικτούς στόχους. Κάποια στοιχεία τα οποία και κάποιες παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, για θέματα τα οποία στην Λευκή Βίβλο χρήζουν ε, πιο λεπτομερούς αντιμετώπισης. Δηλαδή χρειάζονται μέτρα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο θέμα αρμοδιότητας, γιατί υπάρχει και η επικουρικότητα στο σημείο αυτό εδώ. Ε, τα θέματα μεταφορών αντιμετωπίζονται σε πολλά επίπεδα και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Και δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γκρός ότι θα πρέπει να έχουμε σαφέστερους στόχους ε, ε, στην κοινοβουλευτική έκθεση διότι εάν χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε κάτι με το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε είτε σαν νομοθετικό κείμενο είτε σαν ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη θέλουμε ένα κείμενο εφικτό και συνεκτικό Τώρα, για κάποιες πιο πρακτικές παρατηρήσεις, Πρόεδρε. Όσον αφορά το πρόγραμμα 10-10, ε, και άλλοι το είπανε κιόλας, πρέπει να έχουμε πιο περιορισμένους στόχους, λόγω ακριβώς και του οικονομικού κλίματος. Δεν, ε, δεν υπάρχουν χρήματα για να χρηματοδοτήσουν αυτά τα μεγαλοπρεπή σχέδια. χρειαζόμαστε άμεσα αποτελέσματα, ακόμα και για τα net, ε, για τα ten, συγγνώμη, ε, ας πούμε η κατάργηση των σημείων συμφόρενσης. Θα πρέπει να δούμε τους περιορισμένους πόρους που έχουν στη διάθεσή μας, πώς μπορούμε ε, να τους επενδύσουμε καλύτερα. Παραδείγματο χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ πετυχημένο το σχέδιο για την ασφαλή στάθμευση των φορτηγών για να ολοκληρώσω πρόεδρε αυτό το προσπαθώ να πω και προσπαθώ να κάνω μέσω των τροπολογιών που υπέβαλα είναι να επανέλθουμε στα, στις παρατηρήσεις του κ. Γκρόση για τους στόχους θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και να μην προχωρήσουμε με αυτές τις νεφελώδεις ιδέες που είναι ωραίες μεν αλλά δεν έχουν πρακτικό αποτέλεσμα δε Κράμερ, εγώ θέλω και εγώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον εισηγητή για την έκθεσή του Φυσικά είναι πολύ σημαντικά τα θέματα της, ε, των μεταφορών και παίζει εκεί μεγάλο ρόλο η λευκή αυτή βίβλος. Χωρίς μια αλλαγή του τρόπου διακίνησης δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε για να δώσουμε τα παιδιά μας σε κάποιες προοπτικές ζωής. Νομίζω ότι οι μεταφορές στην Ευρώπη εξακολουθούν να είναι πολύ φθηνές Όλα αυτά τα οποία προστατεύουν το περιβάλλον είναι πολύ ακριβά και αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο στην Ευρώπη που δίνει τα λάθο μηνύματα και τη λάθο κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να το τροποιήσουμε. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό <clears throat> το ότι αναφέρθηκε στις πόλεις ο Ματιέ. Γιατί κατά 30% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρωπου στην Ευρώπη ευθύνεται η κυκλοφορία. Έχει ανέβει 35% το ποσοστό των εκπομπών από τις ε, μεταφορές, δηλαδή όλα αυτά τα οποία γίνονται με την, ε, τις προσπάθειες στη βιομηχανία για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, καταστρέφονται και αντιστρέφονται από τι ε, τις μεταφορές. 70% λοιπόν είναι οι, τις μεταφορές είναι οι εκπομπές από τα μεταφορικά οχήματα στις πόλεις. Αυτά είναι τα στοιχεία των ευρωπαϊκών φορέων. Βλέπετε λοιπόν στον τομέα αυτό που υπάρχει πραγματικά το πρόβλημα. Είναι στην οδική κυκλοφορία. Θα σας παραθέσω αυτά που είπε ο δήμαρχος του, του Μονάχου, ο κύριος Φόγκελ, ο οποίος ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία και τόνισε ότι ότι αν συνεχίσει αυτή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων με αυτόν τον τρόπο, στο τέλος δεν θα μπορούμε να πάμε να κουνηθούμε ρούπι. Αυτό το 1971 το είπε. Κανεί δεν κατάλαβε τι εννοούσε τότε. Πρέπει να τροποποιήσουμε λοιπόν τον τρόπο μεταφοράς και κινητικότητας τη πόλη μας. Δεν μπορούμε πια να υποστηρίζουμε τρόπους μεταφοράς που ε, καταστρέφουν ουσιαστικά τι πόλει και χωρί να μιλήσω καθόλου για, τα, για την κλιματική αλλαγή και τα προβλήματά της το Βερολίνο έχει καταστραφεί πολύ περισσότερο από την οδική κυκλοφορία από ότι από τις βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άμα δείτε φωτογραφίες θα το καταλάβετε αυτό και δεν μιλάω καθόλου για την κλιματική αλλαγή ακόμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη σωστή κατεύθυνση στη χρηματοδότηση. 60% όλων των χρημάτων που πηγαίνουν στην Ευρώπη αφορούν τις οδικές μεταφορές, μόνο 20% στους σιδηροδρόμους. Και γι' αυτό έχουμε καταθέσει τροπολογίε, γιατί εκεί πρέπει να αλλάξει αυτή η ισορροπία. Γιατί πάντα εμεί επενδύουμε προ τη λάθο κατεύθυνση. Και μετά μα κάνει εντύπωση ότι δεν πετυχαίνουμε του στόχου που έχουμε θέσει στον εαυτό μα. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι, Ματιέ, αναφέρθηκε και πάλι ποιοι είναι οι στόχοι μείωση για του διάφορου τομεί. Εμεί υποστηρίζουμε να πούμε ότι γενικά οι μεταφορέ θα πρέπει να μειωθούν κατά 30% μέχρι το 2020, γιατί αυτό είναι απαραίτητο Όχι βέβαια μονάχα για να επιτευχθούν οι στόχοι πολύ γρήγορα και μετά ποιος ξέρει τι θα γίνει. Μας ενδιαφέρει όμως να μειώσουμε τη μεγάλη αύξηση που έχει υπάρξει στις μεταφορές και να προσπαθήσουμε να αναστρέψουμε αυτή την ανάπτυξη που υπάρχει. Το 30% αυτό όμως πώς θα γίνει από τα κράτη-μέλη είναι δική τους υπόθεση, αλλά αυτό το 30% για τη μείωση των μεταφορών είναι σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό με έναν τρόπο ο οποίο δεν είναι μεμονωμένο στο κάθε κράτο όπω θέλει. Θα πρέπει να υπάρχει ένα γενικό φορέα ο οποίο αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά. Επίση, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό dumping. Πρέπει να υπάρχει κατά κατατομή μια συλλογική σύμβαση, μια συμφωνία, ώστε να μην υπάρξει το κοινωνικό αυτό dumping και να μην εμποδίσει τι προσπαθίε μα. Είναι πάρα πολλά πράγματα για τα οποία έχουμε ήδη νομοθεσία. Γιατί όμω η Κομισιόν η οποία δεν εξασφαλίσει ότι θα εφαρμόζονται. Όταν έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα στα κάτι μελη η Κομισιόν δεν πιέζει να τα εφαρμόσουν. Είναι απαραίτητο να υπάρξει λοιπόν συνεργασία και με τα κράτη-μέλη. Και το τελευταίο που αναφέρθηκε, ματιά για την ηλεκτροκίνηση στις πόλεις. Αυτό υπάρχει, δηλαδή υπήρχαν ήδη από το 1902 ηλεκτρικά τραμ στο Βερολίνο. Υπάρχουν πέντε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με στις, στις ε, κινήσεις που ένα από αυτά λύνει η ηλεκτροκίνηση. Δεν αντιμετωπίζει τα ατυχήματα, δεν αντιμετωπίζει το θόρυβο, δεν αντιμετωπίζει τη χρήση του εδάφους από, από το από τους δρόμους, ούτε το κόστος για τον καταναλωτή. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν επαρκείς στόχους για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην, ε, στη Γερμανία είπε ότι μπορούμε με χρησιμοποίηση υλικών που υπάρχουν ήδη στην αγορά να μειώσουμε τις εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου. Είναι στα 77 γραμμάρια στο χιλιόμετρο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατά μέσον όρο. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει μηδενίσει όλα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε λοιπόν να θέσουμε στόχους, αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει οι μηχανικοί να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι μονόδρομος η ηλεκτροκίνηση. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε και άλλους τρόπους για να εξασφαλίσουμε την ε, επίτευξη αυτών των στόχων. Χτυπάει το σφυρί του ο πρόεδρος, οπότε σταματάω και σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις των σκιωδών. Ξεκινάμε με τον κύριο Ντεγκράντες Πασκουάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ κάπου παραγνωρίζουμε το τι σημαίνει η Λευκή Βίβλος. Δεν ξέρω αν είναι ένα από τα δώρα των μάγων ή κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι είναι ένας κατάλογος καλών προθέσεων, αλλά παρόλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε την άποψή μας. Νομίζω ότι ο κύριος Γκρός τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ισορροπία και αντιμετώπισε με μια ισορροπημένη προσέγγιση αυτή την έκθεση και έτσι κι αλλιώς δεν τον ζηλεύω. Ξέρει ότι μπροστά του ο κύριος Γκρός έχει την υποστήριξή μας, ξέρει ότι οι τροπολογίες μας θα αφορούν αποχρώσεις, θα είναι συμπληρώματα αυτών που θέλει αυτός να πετύχει. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πραγματικό τέλμα με 413 τροπολογίες από το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο να βγει κανείς. Κάτι για τις τροπολογίες τώρα και στις γενικές γραμμές. Σε ορισμένε χώρες, κύριε και κύριοι, οι οδικές μεταφορές είναι κάτι που δεν είναι απλώς μια επιλογή ή μια λανθασμένη έξι, είναι μια υποχρέωση, διότι δεν υπάρχει καμιά άλλη δυνατότητα. Ο στόχος των διευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να είναι να διασυνδέσει τα εθνικά δίκτυα. Και σίγουρα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι διαπεριφερειακές συνδέσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει φιλελευθεροποίηση των συνδεδρόμων αν δεν υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Η πολιτική για τις μεταφορές θα πρέπει να υποστηρίξει την ενιαία αγορά. Αν δεν έχουμε μία υποδομή ενιαία ευρωπαϊκή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό ο ελεύθερο ανταγωνισμό χωρίς να υπάρχει μία εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστου ή μία εναρμόνιση στο φορολογικό τομέα. Νομίζω ότι αυτά τα οποία θα προκύψουν από την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστου θα πρέπει να βοηθήσουν τι μορφέ μεταφορών που, από τι οποίε προέρχεται αυτό το κόστο. Είναι απόλυτα δυνατόν να μειώσουμε, να διατηρήσουμε το χρόνο ανάπαυση των ε, εργαζομένων και επίσης θα πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση τη ενέργεια ασφάλεια. Όλε αυτέ οι ιδέε σα τι δίνω λιγάκι ε, ακατέργαστες. Όλες αυτές είναι τροπολογίε οι οποίε, περιέχονται, είναι ιδέε που περιέχονται στι τροπολογίε μα και μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο. Για τι άλλε τροπολογίε, κύριε Πρόεδρε με κάθε ε, συντομία θα ήθελα να πω τα εξή. Εμένα δεν μου αρέσουν οι τροπολογίε οι οποίε θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μετακύληση του όγκου μεταφορών από ένα τομέα μεταφορών σε ένα άλλο. Ή αυτοί που θέλουν ότι πρέπει να υπάρξει ευρωβινιέτα σε όλα τα κρατημέλη υποχρεωτικά. Δεν μου αρέσουν αυτέ οι οποίε αφορούν, αφαιρούν τη σημασία τη διαμεθοριακή των ευρωπαϊκών δικτύων και αυτέ οι οποίε θέτουν προσκόμματα για την καλύτερη λειτουργία των αγορών σε κάθε συγκεκριμένο τομέα μεταφορών. Όλα αυτά είναι αξιολογικέ κρίσει, μπορώ να τι σεβαστώ βέβαια, αλλά εμεί θέλουμε να τονίσουμε ότι θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να είναι συνεκτικά με τι απόψει που έχουμε διατυπώσει στο παρελθόν στην Επιτροπή μα. Εγώ πιστεύω με κάθε ειλικρίνεια ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση και να έχουμε ένα σχέδιο έκθεση το οποίο να δείχνει μια επικοδομητική και προοδευτική άποψη σε σχέση με την Ευρώπη και σίγουρα έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον ε, εισηγητή και είναι δεδομένο θα έχει την υποστήριξή μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Αλκαντράουι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες. Θα ζητήσω όμως και από το συγητή να προχωρήσει σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες προκειμένου να καταφέρουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρώτον, θέλουμε έναν ευρύ, ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως και χρηματοδότηση για τον χώρο αυτό. Επίσης, τίθεται και το ζήτημα της καλύτερης διασύνδεσης ανάμεσα στους διάφορους τρόπους μεταφοράς, τα διάφορα μέσα μεταφοράς. Μια καλύτερη διατροπικότητα, λοιπόν, αλλά και καλύτερη διασύνδεση ακόμα και στα πλαίσια του ίδιου τρόπου μεταφοράς. Νομίζω πλέον ότι οι τεχνολογικές γνώσεις που διαθέτουμε μας επιτρέπουν να, να σημειώσουμε πολύ σημαντική πρόοδο. Κάθε φορά που μιλάμε για τις επιπτώσεις στην αγορά, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το άνοιγμα της αγοράς κινείται με την δημιουργία μιας ενό ισότιμου περιβάλλοντο και ενό ισότιμου όχι μόνο ανταγωνιστικού αλλά και κοινωνικού περιβάλλοντο. Θέτω το ακόλουθο ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε τα πράγματα λίγο πιο βραχυπρόθεσμα. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη η κατάσταση. Θα ήταν πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αναλύσουμε συγκεκριμένα τις επιπτώσεις από το πρόγραμμα και να καταφέρουμε να δούμε σε ποια σημεία θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την πρόταση. Δεύτερον, θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε περίπτωση να βρεθούμε σε κάποιο αδιέξοδο, σε κάποιο τέλμα. Σαφώς οι μεταφορές θα αυξηθούν στο μέλλον αν δεν αναλάβουμε τις συγκεκριμένε πρωτοβουλίες που πρέπει να λάβουμε, αν δεν καταβάλουμε προσπάθειες, θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη θέση. Ενδεχομένως να πρέπει να αναλάβουμε δύσκολα μέτρα και θα πρέπει βέβαια να συμπεριλάβουμε και την εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους. Αποτελεί και αυτό μέρος της λύσης. έχουμε και τους περίφημους στόχους για το modal shift, τις αλλαγές στα μέσα μεταφοράς, όχι μόνο για τις μικρές αλλά και τις μεγάλες αποστάσεις. Και στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση δηλαδή, των μεγάλων αποστάσεων, μπορεί τα κέρδη να είναι πολύ μεγαλύτερα, τα ωφέλη από το εγχείρημα. Και θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερες λύσεις όσον αφορά και τις εσωτερικές πλωτές δεν θα πρέπει απλώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λέμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να ελοποιούμε τελικά και τις ε, θεωρητικές μας αυτές τοποθετήσεις. Και ως προς αυτό θεωρώ ότι δεν έχουμε δείξει ιδιαίτερα, ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία αντιστέκονται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αστική κινητικότητα. Πριν από δύο-τρία χρόνια είχαμε ένα σχέδιο δράσης, το εγκρίναμε εδώ πέρα, το πρότεινε προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε στη συνέχεια και ουσιαστικά προέβλεπε μία ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με όλες τις αστικές περιοχές. Στην πράξη όμως τι έγινε. Και υφίστανται ακόμα κάποια πράγματα τα οποία κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία. Κυρία Μπιλπάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει και θα καταβάλει και στη συνέχεια. Είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό έγγραφο. Εν καιρό θα ήθελα να πω καταρχήν ότι συμφωνώ και συμμερίζομαι απόλυτα αυτά που είπε η συντονίστρια μας η κυρία Μέισνα και θεωρώ ότι οι τροπολογίες οι οποίες έχουν παρουσιαστεί από μένα έχουν σαν στόχο κυρίως το να δημιουργηθεί ένα πραγματικό ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αυτό πρέπει να είναι προφανέ. Με τι τροπολογίε αυτό το οποίο θέλω είναι να συμβάλλω στο να εξαλειφθούν όλα αυτά τα προσκόμματα και οι φραγμοί μεταξύ των διαφόρων μορφών μεταφορών, να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα για όλε τι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να οικοδομήσουμε την εδαφική συνοχή η οποία ακόμα ελείπει στην Ευρώπη, ώστε να αναπτύξουμε περισσότερο την ανταγωνιστικότητά μα σε πολλές από τις τροπολογίες υπάρχει μια ιδιαίτερη μνήμα στα σε αυτού που έχουν προβλήματα κινητικά, όχι μόνο γιατί εμεί έχουμε φέρει στην Επιτροπή αυτή διάφορε πρωτοβουλίε και έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα αυτό, αλλά γιατί πιστεύω επίση ότι πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και να συνδέσουμε όλε τι πρωτοβουλίε οι οποίε στο παρελθόν έχουν εγκριθεί από αυτό το Κοινοβούλιο προ την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο να ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα το δικαίωμα των επιβατών και των ατόμων που έχουν προβλήματα κινητικά να υποστηριχθούν από καινοτόμα προγράμματα τα οποία θα δημιουργήσουν ε, θέσεις απασχόλησης και θα δώσουν και μια καλύτερη κατάρτιση για τα άτομα με αναπηρίες γιατί νομίζω ότι στους τομείς αυτούς που υπάρχουν ε, οι καινοτόμες αυτές πρωτοβουλίες μπορούν να απασχοληθούν σε συνθήκες απόλυτης ισότητας με άλλα άτομα στην κοινωνία μας. Πιστεύω ότι αυτό λοιπόν συμβάλλει στη συνεκτικότητα του εγχειρήματό μας. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και στα ευρωομόλογα που είναι ένας πόρος ο οποίος μπορεί να προωθήσει τις υποδομές. Αυτό τόνισε και ο πρώτο Παρόσο στην, τελευταία, στην πρόσφατη Ολομέλεια. Αυτή την κατεύθυνση είχε ο λόγο του. Πρέπει λοιπόν να τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά και να τα ενσωματώσουμε σε μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και τι περιφερειακές τοπικέ αρχέ, που ακόμα και αν αντιστεκόμαστε πολλέ φορέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν πραγματικά ένα σημαντικό ρόλο και σημαντικέ αρμοδιότητε στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να βρούμε τρόπου να ενσωματώσουμε και τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ και να οικοδομήσουμε μια λήψη αποφάσεων με μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω γιατί αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Όπως αναφέρθηκε και ο εισηγητής, πρέπει να μιλήσουμε και για τις υπεριφερειακές περιοχές και τα νησιά. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία βρίσκονται στις τροπολογίες μου έχουν σαν στόχο να τροποποιήσουν και τις ε, συνθήκες ε, <clears throat> εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών και την χρήση των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται στα δημόσια έργα. Μέσα σε μια εποχή κρίσης, οι τροποποιήσεις που έχουν ε, εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να αφαιρέσουν την ε, ευελιξία στον τομέα αυτά. Τουλάχιστον θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη τις διαμαρτυρίες του κλάδου για τις ε, αποφάσεις αυτές. Πιστεύω επίση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο καινοτομία για τι μεταφορέ, γιατί αυτό θα είναι σύμμορφο και στην ίδια κατεύθυνση με την Ευρώπη 2020 που είναι μια από τι στρατηγικέ μα γραμμέ και κάτι τέτοιο θα μα επιτρέψει να αναπτύξουμε με πιο βιώσιμο και πιο αποτελεσματικό τρόπο τι προσπαθειέ μα και να δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία που είναι κάτι που οπωσδήποτε χρειαζόμαστε στο μέλλον. Χρειάζεται επίση ειδική ρύθμιση για τα οχήματα αναψυχή. Αυτό είναι ένα τομέα σε άνθηση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τα οχήματα αναψυχή και σε μένα μου έρχονται συνέχεια αιτήσει και ερωτήματα σε σχέση με αυτά τα οχήματα. Η μπλε ζώνη τώρα που αναφέρεται είναι μια πρόταση, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να τη συνδυάσουμε με την πρόταση για, τους, για τις λεωφόρους της θάλασσας. Και πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο, ο θαλάσσιος τομέας, ο τομέας των ναυτικών μεταφορών είναι στρατηγικός και να υποστηρίξουμε προγράμματα καινοτομία στον τομέα αυτό που θα μας επιτρέψουν ο ευρωπαϊκός <clears throat> ναυτικός τομέας να βγει από την κρίση στην οποία βρίσκεται με την μεγάλη με το μεγάλο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει από την Νοτιοατολική Ασία και να παίξουμε και ένα πρωτοπόρο ρόλο ως Ευρώπη των μεταφορών με μείωση των εκπομπών, με ενεργειακή αποδοτικότητα και με προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε εγκρίνει σήμερα μία σειρά από τροπολογίε της ΕΜΣΑ. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, λύσεις που προτείνει για την αντιμετώπιση παραγωγικά της πειρατείας, να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ε, εναρμόνιση στις ε, αστικές συγκοινωνίες και να λάβουμε υπόψη και την δυνατότητα να αναπτυχθεί η μεταφορά με τραμ. Πάντα όμως μέσα στα πλαίσια της επικορικότητας της Ευρωπαϊκής Πόλης. Είναι απαραίτητο να δώσουμε μια αποφασιστική υποστήριξη στα διευρωπαϊκά σχέδια μεταφορών με μια σαφή διατύπωση ορισμών του τι είναι αυτό που θέλουμε και ελπίζω ότι όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια καλύτερη προσβασιμότητα, μια καλύτερη εδαφική συνοχή και όλα αυτά θα οδηγήσουν στην ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία λέχθηκαν ήδη. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να τα εξάρω εδώ. Πρώτα απ' όλα οι κοινωνικές συνθήκες. Νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκρός, ο οποίος τόνισε τη σημασία αυτών των κοινωνικών συνθήκων και εμείς φυσικά δεν τις θέτουμε ένα αμφιβόλο. Είναι αυτή τη στιγμή ένα τομέα ο οποίος έχει ένα πρόβλημα image, εικόνας. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι η κατάρτιση και η περιττέρω εξειδίκευση των εργαζομένων θα είναι σημαντική, γιατί χρειάζεται να υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό στις μεταφορές και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα με μία ε, μείωση των κοινωνικών προδιαγραφών, αλλά αντίθετα μόνο με την καλύτερη κατάρτιση. Από την άλλη πλευρά θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη βελτίωση στις διαμεθοριακές ε, συγκοινωνίες. Αυτό δεν αφορά μονάχα τον οδικό τομέα και δεν αφορά μονάχα την ε, διευκόλυνση και την απλοποίηση των ε, ελέγχων. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε και τα σημεία συμφόρησης στις υποδομές και την συσσόρευση των υπερβολικών κανόνων. Εδώ μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη βελτίωση. Επίση, η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι σημαντική να μειώσουμε την ένταση εργασίας στις μεταφορές. Αυτό είναι μια απόλυτη αναγκαιότητα. Μπορούμε με καλύτερη αποδοτικότητα να λειτουργήσουμε καλύτερα τις μεταφορές και να αποφύγουμε την μεταφορά, μάλλον την κίνηση κενών οχημάτων ώστε να μην υπάρχουν περιττές κινήσεις οχημάτων. Όλα αυτά με μια εναρμόνιση η οποία θα εξασφαλίσει την ε, εφαρμογή αυτών των κανόνων. Και η ασφάλεια είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα μέρημνας για μένα και εδώ είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν περισσότερο χρόνο ανάπαυσης οι οδηγοί των φορτηγών και αυτό να αντιμετωπιστεί όχι μονάχα υπό την οπτική γωνία των συνθηκών εργασίας αλλά και σε ό,τι αφορά την ίδια την οδική ασφάλεια. Γιατί πολλές φορές οι οδηγοί είναι και αυτοί υποχρεωμένοι να κοιμούνται στην άκρη του δρόμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται βελτίωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Τικάου. Θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να συγχαρώ τον κύριο Γκρόσο τον υποστηρίζουμε πλήρως και ελπίζω ότι θα στεφθούν και με επιτυχία οι συμβαστικές τροπολογίες. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και την Κομισιόν για αυτή την Λευκή Βίβλο. Είναι ένα πλήρες έγγραφο το οποίο συμπεριλαμβάνει πολλά μέτρα και εκφράζει την δέσμευση της Κομισιόν ε, και για την, τα νομοθετικά διαβήματα τα οποία απαιτούνται αλλά και τα μέτρα τα οποία θα υιοθετήσει στο μέλλον. Ε, υπέβαλα κάποιες τροπολογίες ε, γιατί θέλουμε στα, στα, στα επόμενα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια να ληφθεί υπόψη και η, το, η κατάσταση της κυκλοφορίας στις νέες χώρες. Θα πρέπει δηλαδή με κάποιο τρόπο να ε, καλυφθεί το κενό που υπάρχει ανάμεσα στις νέες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις, ε, και τις υπόλοιπες θα πρέπει, ε, αναφέρεται, ε, να αυξηθεί και ο αριθμός ε, θέσεων στάθμευσης των φορτηγών που πρέπει και να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια αλλά και υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία χρήζουν βελτίωση. παραδείγματος χάρη στον σιδηροδρομικό τομέα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα δίκτυο ταχείας κυκλοφορίας στο σιδηροδρόμων που να ενώνει όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Επίσης, αναφέρθηκα στο πρόγραμμα NIAD. Θέλουμε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τα εσωτερικά ύδατα. Μια παρόμοια πολιτική δηλαδή για τα εσωτερικά ύδατα όπως για την, για την θάλασσα. Θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας και και τα ποτάμια και τις άλλες πλωτές οδούς της, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προωθήσουμε επίσης και τις υποδομές για την προώθηση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο ε, να παίρνει από, την, από την Κομισιό κάθε πέντε χρόνια ένα μια σειρά μέτρων ε, που θα υιοθετεί για την ε, υλοποίηση των, ε, των στόχων μας. Θα πρέπει κάθε πέντε χρόνια η Κομισιόν να συνερώνει την πρόοδο. Ευχαριστώ κύριε Στρομόσα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα λεπτό θα μιλήσω. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Τρία σημεία θέλω να θίξω γιατί 30 τροπολογίες έχω υποβάλει. Αναφέρεστε στον τομέα των logistics και δίνετε κάποια αριθμητικά δεδομένα. Θεωρώ ότι το τομέας αυτός είναι πιο σημαντικός από ό,τι λέτε εσείς. Ο τομέας της, των logistics είναι ο τομέας αυτός, ο οποίος αν δεν λειτουργεί σωστά επηρεάζεται όλη η ευρωπαϊκή οικονομία όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Αν πρέπει λοιπόν να κάνουμε πιο ευέλικτους κάποιους δείκτες ε, στη λευκή αυτή βίβλο, προκειμένου να προστατεύσουμε την κερδοφορία του τομέα των logistics, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεύτερον, μία από τις τροπολογίες μου που θεωρώ σημαντική έχει να κάνει με την ε, εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους τη διεθνή εσωτερική του εξωτερικού κόστους. Νομίζω ότι για όλα τα μέσα μεταφοράς και για, τον, και για τη μεταφορά επιβατών και για τις εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να γίνει αυτή η εσωτερική του εξωτερικού κόστους. Συμφωνώ με, τα, με, όσα, με όλα όσα λέγονται για τα TNT. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αντισταθούμε, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αντίσταση κάποιων κρατών μελών. Θα πρέπει τα μέτρα αυτά τα οποία επιφέρουν θέμενη αξία να είναι υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τις σιδηροδρομικές μεταφορές, συμφωνώ με την ιδέα αυτή να έχουμε, μια, να έχουμε ανεξάρτητες εθνικές αρχές επιτήρησης και θα πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει και μια αντίστοιχη Ευρωπαϊκή υπηρεσία επιτήρησης. Θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλές συμβαστικές τροπολογίες. Ο κύριος Κουμουτσάκος έχει το λόγο. Thank you, <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ χαιρετίζω το υψηλό επίπεδο της εργασίας του Ματιού. Νομίζω με την απαραίτητη συνεργασία θα μπορέσουμε να επιτύχουμε στο να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Τόσο και ο κύριος ε, Ματιό όσο και άλλοι αναφέρθηκαν σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν μέτρα τα οποία να είναι εφικτά και ρεαλιστικά. Αυτός πρέπει να είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος του έργου μας. Μέχρι ότου καταλήξουμε στο τελικό κείμενο αυτής της έκθεσης. Του του λεχθέντος. Θα ήθελα να αναφέρω επειδή ακριβώς μιλάμε για αυτή την προσέγγιση που πρέπει να είναι ρεαλιστική, ότι οι περιφερειακοί κανόνε κανόνες και οι περιφερειακές ρυθμίσεις θα πρέπει να αποφευχθούν σε τομείς μεταφορών που έχουν πραγματικά παγκόσμια εμβέλεια όπως είναι η ναυτιλία όπου πάρα πολλά θέματα θεσπίζονται ήδη και διέπονται από διεθνείς συμβάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν συζητούμε εκθέσεις που έχουν να κάνουν με την αυτιλία. Έχω δύο σημεία τα οποία θέλω να τονίσω για τη μείωση του εκπαιδευμένου διοξιδίου του άνθρακος. Είναι γνωστό ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Και η πρόσφατη έγκριση του EIDICMP είναι μια καλή απόδειξη για αυτό το γεγονός. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε μέτρα περιφερειακού χαρακτήρα που, που σε τελική ανάλυση θα αποδειχθούν αντιπαραγωγικά. Ένα δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω σε σχέση με την εναρμόνιση της εκπαίδευσης των ναυτικών με διεθνή πρότυπα μέχρι το 2012 νομίζω ότι για το σημείο αυτό πιστεύω ότι οποιαδήποτε νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ε, ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές όπως είναι οι προδιαγραφές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την εκπαίδευση της βάρδιας κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να μην υπάρξουν πρόσθετες υποχρεώσεις και περιφερειακά μέτρα. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σωστές συμβαστικές λύσεις για διάφορα θέματα και αυτό συμπεριλαμβάνει τα θέματα που έδειξε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και προσβλέπω στη συνεργασία με τον Ματιό και τους υπολείπους συναδέρφους για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Τισέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω χαιρετίζοντας και εξαίροντας το έργο του εισηγητή, το έγγραφο το οποίο μας παρουσίασε και το οποίο νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση συζήτησης. Ο κύριος Δεγκράτες Πασκουάλ είπε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πλαίσιο ε, μέσα στο οποίο υπάρχουν αιτήσει και άμα έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο απαιτήσεων αυτό δεν θα ενισχύσει την συνεκτικότητα του τη εκθέσεώ μα. Ο στόχο του να πετύχουμε μια ενιαία αγορά και ένα ενιαίο χώρο διακίνηση για του πολίτε μα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εξίσου είναι σημαντικό η πολιτική μεταφορών μα να λάβει υπόψη και τι ιδιαιτερότητε των περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διάφορα σημεία συμφόρηση και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι πολίτε σε αυτές τι ε, περιοχές. Έρχομαι από μια υπερπεριφερειακή περιοχή, τη Μαδέρα, όπου τα λιμάνια και τα αεροδρόμια είναι κεφαλαιόδη για να μπορέσει να υπάρχει μια πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και υπάρχει η ανάγκη της συνοχής για την ενιαία αγορά. Χωρίς λιμάνια, χωρίς αεροδρόμια, οι υπερπεριφερειακές ε, περιοχές της Ευρώπης δεν μπορούν να έχουν καμία πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Θέλω λοιπόν να χαιρετήσω το ανοιχτό πνεύμα του κυρίου Γκρός για να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά στην εκθεσή του και θέλω να υπογραμμίσω ακόμα δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει η ανάγκη να αναπτύξουμε ένα κατάλληλο και θετικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί μια πραγματική θαλάσσια οικονομία μέσα από τις λεωφόρους της θαλάσσης που θα πρέπει να αποτελέσουν και τη βάση των θαλασσίων οδών και η βάση για να δημιουργηθούν πλατφόρμες εξέδρες επιμελητίας ουσιαστικά χώροι από τις οποίους θα κανονίζεται η διακίνηση των, των εμπορευμάτων. Αυτό καλύπτεται από διάφορα προγράμματα όπως το Μάρκο αλλά επίσης θα πρέπει να υπάρξει και ανάπτυξη προγραμμάτων για τις θαλάσσιες υπηρεσίες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή που δεν αντιμετωπίζει τις ανάγκες των ε, υπερπεριφερειακών περιοχών και πρέπει να μην λησμονηθούν αυτές οι περιοχές όπως τόνισαν προηγούμενες λευκές βίβλοι και αυτές είναι περιοχές όπου ζει και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεμπάκερ. Thank you, Chair. Um, I would like to thank... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για την φοβερή δουλειά που έχει κάνει και για τις τροπολογίες επίσης που έχουν υποβληθεί και αυτές που θα υποβληθούν. Ε, και εγώ υπέβαλα κάποιες τροπολογίες. Ένα πράγμα το οποίο θέλω να τονίσω είναι το εξή. Η πρόταση της Κομισιόν είναι να εσωτερικευθούν τα εξωτερικά κόστη. Ήθελα να πω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την διπλή φορολογία. Ο τομέα των μεταφορών είναι ανταγωνιστικό τομέα, σημαντικός για τι οικονομίε μας και θα ήθελα να τονίσω το ότι δεν μπορούμε να φορολογήσουμε διπλά τις ε, επιχειρήσεις αυτές. Εμείς, ας πούμε, στα λιμάνια προσπαθούμε να προσελκύσουμε νέες εταιρείες και ε, να αφήσουμε ανοιχτή όσο δυνατόν περισσότερο την μεταφορά ε, προς το εσωτερικό της χώρας από το λιμάνι. Άρα η αρχή της διπλής φορολόγησης είναι πάρα πολύ σημαντική για μας να αποφευχθεί. Επίσης κάτι άλλο ε, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στις, στα στις πλατφόρμες πολυμέσων για τα 20%. Θα, το πρόβλημα δεν είναι η αποτελεσμα, η, ο αριθμός των πλατφόρμων, αλλά η αποδοτικότητά τους, η αποτελεσματικότητά τους. Επίσης, ήθελα να κάνω μία τροπολογία για την πρόταση του, προέδρου, του συγκητή που είπε ότι το 10% των TNT θα πρέπει να προωθηθεί στην αυσιπλοεία ε, εμείς πιστεύουμε ότι ούτως ή άλλως ε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο τεν και τα λιμάνια και τα εσωτερικά λιμάνια κτλ. Βεβαίως ε, προσδοκάμε σε μια απολυτική συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Γέγκερ για την Κομισιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ποιότητα της δουλειάς του και να συγχαρώ όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, για τις 313 τροπολογίες που υπέβαλαν. Πολλές από τις τροπολογίες που εξετάσαμε προσεκτικά δείχνουν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει αλλά και το εύρος των ιδεών ε, για τον ε, τομέα αυτό. Ε, η Κομισιόν πιστεύει ότι η έκθεση Γκρέσ υποστηρίζει ένα φιλόδοξο όραμα για τις μεταφορές. Ελπίζουμε ότι οι πολιτικές μας γενικώ συγκλίνουν και γενικώ η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα ε, θετική για την Κομισιό. Ε, έχουμε όμως κάποιες αντιρρήσεις τις οποίες ε, θα τις αναφέρω, έστω και αν επαναλαμβάνομαι. Η ολοκλήρωση της εταιρικής αγοράς είναι πάρα πολύ σημαντική. Εξού και καλωσορίζουμε την, ε, το τέταρτο συνδρομικό πακέτο μέχρι το τέλος του 2012, όπου θα υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα στην, στους, σε αυτούς που διαχειρίζονται τις τις μεταφορές ε, και ε, ε, τους ρυθμιστές. Καλωσορίζουμε την το Blue Belt, την, την γαλάζια αυτή ζώνη. Απ' την άλλη πλευρά όμως πιστεύω ότι οι κανόνες για την οδήγηση και τον χρόνο ανάπαυσης δεν θα πρέπει να αλλάξουν, απλώς θα πρέπει να γίνεται σωστή εφαρμογή. Επίσης ε, θέλουμε να τονίσουμε ότι στην Λευκή Βίβλο η Κομισιόν έχει θέσει κάποιους στόχους και ενδεικτικούς ε, στόχους για το 2020-2050. Έχουν τεθεί και άλλοι στόχοι για το 2020 μέσα στα πλαίσια ε, του πακέτου ενέργειας και κλίματος και αποτελούν το αποτέλεσμα λεπτομερών μελετών αντικτύπου και έχουν διαμορφωθεί διάφορα σενάρια ούτως ή άλλως οποιαδήποτε βελτίωση των στόχων αυτών είναι ευπρόζεκτη. Όμω, εάν υπάρξουν και άλλοι στόχοι, μπορεί να ε, μην μπορέσουμε να του υλοποιήσουμε, διότι μπορεί να είναι πολύ φιλόδοξοι, να μπορεί να μην ταιριάζουν με τους στόχους που έχουμε ήδη θέσει. Το 2020 είναι σε 9 χρόνια και είναι πολύ κρίσιμη περίοδο και για τι μεταφορέ, αλλά γενικότερα ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση. Άρα η προσθήκη πολλών στόχων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλη την, όλο το πακέτο. Ξέρετε ότι τον Οκτώβρη ε, ε, επικυρώσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τον Ε, Άκουσα πολύ προσεκτικά όλα όσα ακούστηκαν σήμερα, τα υποστηρίζουμε, αλλά θέλουμε και μεγαλύτερη υποστήριξη στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη νέα προσέγγιση. Γιατί αυτά τα δίκτυα ε, στηρίζουν στηρίζονται στην ε, κατάργηση των σημείων συμφόρησης, ε, σε καλύτερη, ε, σε καλύτερη διαχείριση και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων και όχι η εμφάνιση ας πούμε 25 σημείων συμφόρησης. Κάποιοι αναφέρονται στο ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την επίτευξη των στόχων μας. Το ίδιο και η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους. Η η, η, η, η ορθολογική φορολογική πολιτική. Αυτά βοηθάνε. Όπως είπε και ο κύριος ε, Γκρόσο, η Λευκή Βίβλος περιγράφει ένα σενάριο το οποίο προβλέπει κάποιες μεταφορές για τις αποστάσεις ε, των benchmark, ε, τα 400 χιλιόμετρα που αναφέρονται για, του για τους σιδηροδρόμους και τα σιδερικά ύδατα σε σχέση με τις οδικές μεταφορές δεν είναι ε, ένας στόχος αυτός καθεαυτός, δεν είναι αυτός σκοπός μάλλον, είναι ένας στόχος, επιθυμητός στόχος. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της Κομισιόν για όλες τις ε, ε, τροπολογίες ε, που υπευλήθηκαν θα ήθελα να να αναφέρω ε, κάποιες τροπολογίες οι οποίες μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Είναι σαν διαγωνισμός καλονής. Δεν μπορώ να τους να αναφέρω όλες τις, ε, τις τροπολογίες που θα θέλαμε, αλλά αυτές οι πέντε μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. 205, 121, 84, 91 και 110. Ε, κύριε Γκρός, έχετε πάλι το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδελφούς για τη συμβολή τους. Νομίζω ότι θα έχετε κατανόηση αν δεν απαντήσω λεπτομεριακά σε όλα αυτά τα οποία ελέγχθηκαν. Όλα αυτά που είπατε τα έχω καταγράψει εδώ πέρα. Δεν πρέπει να ανησυχείτε. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να μην τα πούμε όλα, αλλά από την άλλη πλευρά να εξασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών που θέλουμε να επιτύχουμε και μια ισορροπία μεταξύ του ρεαλισμού και της απαραίτητης πίεσης που πρέπει να ασκηθεί γιατί δεν μπορεί να έχει κανείς και ρεαλισμό και να προωθεί τα πράγματα προς τα εμπρός. Για την Κομισιόν εγώ συμφωνώ με τους στόχους τους οποίους αναφέρει η Κομισιόν, τους ευρύτερους στόχους. Ίσως είναι κάτι το οποίο βασίζεται και στην ηλικία μου, ότι πρέπει να δούμε πρώτα τι γίνεται στα επόμενα δέκα χρόνια και μετά τι θα γίνει αργότερα. Είναι απαραίτητο Επομένως μπορεί κανείς να το δει αυτό σαν μια μορφή ρεαλισμού αν θέλετε. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πολύ καλές τροπολογίες οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Η προθεσμία για τις τροπολογίες καταρχήν 22 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε και στις ε, 22 Νοεμβρίου τροπολογίες και 20 Δεκεμβρίου είναι οι ψηφοφορίες στην Επιτροπή μας. Ακολουθούν τα θέματα φορολογίας ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας και έχει, είναι συντάκτρια της νομοδότησης η κυρία Σαμπίνε Βίλς. Αγαπητοί και αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εγώ υποστηρίζω ε, βασικά την πρόταση της Κομισιόν η οποία έχει μια γενική κατεύθυνση η οποία μπορεί να μα επιτρέψει να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση όλων των ενεργειακών πηγών μέσα από ένα τεχνικά ουδέτερο πλαίσιο αλλά συγχρόνω, να δημιουργηθεί και μια μορφή, μια σειρά κινήτρων ώστε να υποστηριχθεί η παραγωγή ενέργειας που οδηγεί σε μικρότερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Είναι, κύρια, είναι τρία τα κύρια φορολογικά κριτήρια κίνητρα τα οποία αναφέρονται γιατί αναφέρουν την ε, μείωση του διοξιδίου του άνθρακος, εξοικονόμηση ενέργειας και επίσης αύξηση της αποδοτικότητος της χρησιμοποίησης ενέργειας και οικολογικότερη παραγωγή ενέργειας. Δυστυχώς, εξακολουθεί να υπάρχει η απαγόρευση της φορολογίας των καυσίμων στα, στα αεροπλάνα και στα πλοία κάτι για το οποίο δεν υπάρχει ακόμα μια πραγματική αιτιολόγηση. Η Κομισιόν έχει συμφωνήσει με το Συμβούλιο για το να ξεπεραστεί αυτή η απαγόρευση στην επόμενη φορά που θα αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία. Το γεγονός ότι το 2012 ε, θα τεθεί σε λειτουργία και το σύστημα εκπομπών διοξιδίου του Άνθρωπος και για τις αεροπορικές ε, συγκοινωνίες δεν δικαιολογεί μια καθυστέρηση στο, στη φορολογήση αυτών των μορφών μεταφοράς, των καυσίμων για τα πλοία και τα αεροπλάνα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να καταλάβουμε αν μπορεί να βρεθεί μια λύση η οποία θα βασιστεί σε επικουρικότητα αλλά θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να φορολογούν σε, στα τα καύσιμα για, τα, για τις και αεροπορικές συγκοινωνίες. Υπάρχει η δυνατότητα να διευρυνθεί αυτή η βάση και με το να αναφέρεται σαφώς στα, στο κόστος των εισιτηρίων. Υπάρχουν επίσης πολλά κράτη τα οποία έχουν κάνει συμφωνίες για αμοιβαία ε, ρύθμιση φορολόγησης για να αποφύγουν προβλήματα ανταγωνισμού. Η συμφωνία του Σικάγο, του, δεν έχει στο περιεχόμενό τους καμία απόφαση για την ε, ε, απαγόρευση φορολογίας στα αεροπορικά καύσιμα, απλώς μόνο τα καύσιμα τα οποία βρίσκονται ήδη στα αεροπλάνα. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια καλύτερη ρύθμιση για να εσωτερικοποιηθεί και το εξωτερικό κόστος στις θαλάσσιες μεταφορές. Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε σωστέ συνθήκε ανταγωνισμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, θα πρέπει να γίνει ένα πρώτο βήμα προ την κατεύθυνση αυτή οι προτάσεις αυτές δεν θα είναι μια μεγάλη τομή, αλλά θα είναι τουλάχιστον ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς ένα πιο βιώσιμο και αηφόρο σύστημα μεταφορών. Θέλω εγώ να υπογραμμίσω ιδιαίτερα τις ε, εξαιρέσεις που προτείνει η Κομισιόν, ώστε η ενέργεια που παράγεται από τα πλοία στα λιμάνια δεν καλύπτεται από τις απαγορεύσεις αυτές φορολογίες. Και αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται και στην, στους εσωτερικούς, αυσιπλοεία σε εσωτερικούς υδάτινους δρόμους και περιμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί από τις 10.30 ω 11.30 θα συζητήσω με τους πιο συζητητές για τα περαιτέρω. Κάντσια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να εκφράσω κάποιες απορίες όσον αφορά αυτή την οδηγία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια βέβαια και ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες θα καταφέρουμε να ανταλλάξουμε και κάποιες απόψεις. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την πρόταση Κομισιόν, διότι Ούτως ή άλλως η οδηγία είχε σαν στόχο να ισορροπήσει εκ νέου την αγορά. Όμω, εάν σκεφτούμε ότι αυτή η οδηγία προβλέπει μία αύξηση των ε, συντελεστών, ε, των συντελεστών των φορολογικών ε, που εφαρμόζονται στα διάφορα ενεργειακά προϊόντα για τα 6-7 χρόνια, εάν εφαρμοστούν, θα έχουν μια αύξηση 400% για τα καύσιμα αυτά. Με τον τρόπο αυτό και αφαιρείται και το πλεονέκτημα που θα είχαν ε, τα κράτη-μέλη, τα οποία θα τους, ε, πλεονέκτημα το οποίο θα το είχαν μέχρι το 2023. Λοιπόν, πιστεύω ότι τα, τα, προϊόντα αυτά ε, ήδη έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και πιστεύω ότι αυτό το μέτρο το οποίο προβλέπετε εδώ είναι λάθος. Θα έπρεπε να το επανεξετάσουμε. Ίσως για το επαγγελματικό ντίζελ θα έπρεπε να έχουμε μια πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση, κυρίως το ντίζελ που ε, χρησιμεύει για τις οδικές μεταφορές. Έχουμε Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες για να αντικαταστήσουμε ε, το, το πάρκο των φορτηγών, των μεταφορικών μέσων τέλος πάντων. Λοιπόν, εάν θεωρήσουμε ε, τον, ε, αν εξετάσουμε μάλλον τον κλάδο αυτών της, της βιομηχανίας μας, ε, το ντίζελ είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, μπορούσε, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία αυτή για να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας στις αναπτυσσόμενες αγορές. Το, ο συντελεστής φορολογίας που επιβάλλεται εδώ θα οδηγούσε στην εξαφάνιση των καυσίμων που έχουν λιγότερο αντίκτυπο όσον αφορά την στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα, τα καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα, ε, η στάση μας θα πρέπει να επανεξεταστεί έτσι ώστε να μην ε, εξαφανιστούν. Ευχαριστώ κύριε Τιμπάκα. Ο κύριος Τιμπάκα μάλλον. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εργάζομαι και έχω ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και στη δική μα Επιτροπή και στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Βέβαια, στη συγκεκριμένη αυτή γνωμοδότηση πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε προφανώ στο τμήμα που αφορά τι μεταφορέ. Είναι σωστό αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αυτό που θα πρέπει να στοχεύουμε είναι βιώσιμε μεταφορέ και καλύτερη φορολόγηση των ε, προϊόντων αυτών μολύνουν περισσότερο το περιβάλλον και μία εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην έχουμε πολλά διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα ανά κράτο μέλο. Είναι επίση πολύ σημαντικό να πούμε ότι με την πρόταση αυτή ο στόχος είναι να αλλάξουμε τη στάση των χρηστών, των καταναλωτών, όχι το να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα. Συνεπώς, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να δραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο. Συμφωνώ με τη βασική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε, προβλέπονται εδώ πέρα και κάποιε εξαιρέσει. Και αν θέλουμε όντω να δημιουργήσουμε ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού, θα πρέπει οι ίδιοι κανόνε να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Και για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό να αποφύγουμε όσο το περισσότερο τι παρεκκλήσει και τι εξαιρέσει. Μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι όλα τα κάψιμα θα πρέπει να τυχαίνουν του ίδιου φορολογικού καθεστώτο, μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά τώρα τα βιοκαύσιμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δει πώς θα αντιμετωπίσει τα βιοκαύσιμα, τα οποία πολλέ φορές εξαιρούνται. Επίσης, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια στάση που θα είναι τεχνολογικά ουδέτερη είναι πολύ σημαντικό πάλι διάφορες μορφές τεχνολογίας να τυχαίνουν της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης. Και πραγματικά θέλουμε να προωθήσουμε μια πολιτική καινοτομία, τότε η φορολογική μας πολιτική θα πρέπει να είναι ουδέτερης προς την τεχνολογία. Να ευχαριστήσω το συντάκτη γνωμοδότησης. Συμφωνώ με τα περισσότερα και θα υποβάλω βέβαια και κάποιες τροπολογίες. Και ελπίζω να καταφέρουμε να καταλήξουμε έτσι σε μια καλύτερη πρόταση. Ο κύριος Κράμερ. Κύριος Κράμερ. Πρέπει να δούμε πόσο σοβαρά παίρνει η Κομισιόν και το Συμβούλιο τα θέματα εκπομπής αερίου του θερμοκηπίου. Ξέρουμε ότι στη στρατόσφαιρα είναι πολύ πιο επικίνδυνες οι, οι εκπομπές και 300 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις εναρίες μεταφορές. Κάθε χρόνο αν είχαμε αυτά τα χρήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές θα είχαμε καταφέρει, όπως είπε και η κυρία Τσίκαου, να συνδέσουμε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και θα είχαμε καταφέρει να συνδέσουμε όλες τις διαμεθοριακές συνδέσεις. Αλλά όχι, τα δίνουμε αυτά στη λάθος κατεύθυνση. Όταν μιλάμε για μη φορολόγηση, ουσιαστικά μιλάμε για μία επιδότηση που δίνουμε στις αεροπορικές εταιρείες και επίσης άμα πάρουμε τις μεταφορές στην ανοιχτή θάλασσα καίγεται βγαίνουν διοξίδια του διοξιδίου του άνθρακος και αυτό δημιουργεί περισσότερη ρήπανση η ναυτιλία σε, στην ανοιχτή θάλασσα είναι σαν την καύση απορριμμάτων χωρίς να υπάρχει κανένα φίλτρο. Και αυτή τώρα παίρνει φορολογική ελάφρυνση. Με ποιο δικαίωμα. Και με ποια λογική να μεταφέρουμε προϊόντα τα οποία τα πηγαίνουν από τη Σκανδιναβία στο Μαρόκο, τα επεξεργάζονται στο Μαρόκο και ξαναγυρίζουν στη Στοχόλμη για να σερβιριστούν εκεί. Όλα αυτά γίνονται με τα δικά μας χρήματα, με τα δικά μας χρήματα των φορολογημένων. Εμείς τα φορολογούμε αυτά, διαλύουμε το περιβάλλον και τα πληρώνουμε και είμαστε χαρούμενοι. Θέλω να μας πει κάποια στιγμή η Κομισιόν, σταματάμε πια, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Αν θέλουμε να έχουμε τους σιδηροδρόμους, θα πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει κάποιο περιορισμό στις εκπομπές. Και ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα για τους αυτοκινητοδρόμους και για τα φορτηγά τα οποία ξεπερνούν τους 12 τόνους. Αλλιώς μπορούμε να θέτουμε στόχους 30, 40, οτιδήποτε, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, νίξ. Ποτέ δεν θα φτάσουμε τους στόχους αυτούς. Το μόνο μέτρο που έχει η Κομισιόν είναι η χρηματοδότηση. Αυτό είναι ο μόνο μοχλό που έχει να αντιμετωπίσει την εθνική επικουρικότητα. Άμα δεν τον χρησιμοποιήσει, τον έχει χάσει. Είναι δυνατόν να περιλάβουμε λοιπόν τη φορολογία της κύριοζηνή. Δεν θέλουμε να την φορολογήσουμε επειδή είναι <clears throat> ένα επειδή Θέλουμε να θίξουμε την αεροπορική βιομηχανία. Οποιοδήποτε αεροπλάνο έρχεται στην Ευρώπη και φορτώνει κυροζίνη πρέπει να φορολογείται, πόσο οποιοδήποτε αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει στο βενζινάδικο. Εδώ λοιπόν θα φανεί αν η Κομισιόν, αν το Συμβούλιο, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν πραγματικά να πάρουν μια θαραλέα θέση ή απλώς θέλουν να διατηρήσουν τις επιδοτήσεις αυτές οι οποίες κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση. Αλλά οι επερχόμενες γενιές θα τα θυμηθούν αυτό και θα τα φορτώσουν στην πλάτη μας αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιος και ο μας είπε ήδη ότι δεν μου αρέσει αυτή η οδηγία και ούτε και εμένα μου αρέσει. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος θα προσπαθήσω να εστιάσω την προσοχή μου στις πτυχές που δεν με ικανοποιούν. Αφήνω τι επένδυση για κάποια άλλη στιγμή όταν βελτιωθούν τα πράγματα και πάντα ελπίζω θα γίνει κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά την εξαίρεση του επαγγελματικού ντίζελ, η πρόταση Κομισιόν είναι ε, πληθωριστική και άδικη για τις περιοχές της ε, περιφέρειας. Ένα μέτρο όπως αυτό κυρίε και κύριοι δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να αυξήσει ε, δυσανάλογα το κόστος των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών. 60% του τελικού κόστους είναι το κόστος των καυσίμων στις μεταφορές. Εμείς είμαστε εναντίον ορισμένου μέτρου κατά των ε, οδικών μεταρρυθμίσεων εάν δεν υπάρχει η ελευθερία στη θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά. Επίση, το άρθρο 103 των συνδικών στο οποίο βασίζεται η πρόταση τη η φορολογική εναρμόνιση μπορεί να γίνει μονάχα στο βαθμό στον οποίο αυτή η φορολογική εναρμόνιση είναι απαραίτητη για να μπορέσει να εξασφαλίσει την δημιουργία και τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και να αποφύγει τι τρευλώσει ανταγωνισμού. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτή η προπόθεση γιατί δεν υπάρχει ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων μεταφορά και τρόπων μεταφορά. Όπως σας είπα λοιπόν, η κατάργηση του επαγγελματικού diesel σημαίνει αύξηση του κόστους μεταφορές στις περιφερειακές περιοχές στις και περιφερειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των άλλων. Για τα βιοκαύσιμα επίσης και μη φορολογία τους. Η πρόταση της Κομισιόν είναι συνεκτική με τις αρχές της βιωσιμότητας για την οδηγία που αφορά τις ανανεώσιμες ενέργειες. Αλλά θα πρέπει να καταγράψουμε ότι είμαστε εναντίον αυτών των κριτηρίων που θεωρούμε ότι είναι καταχρηστικού χαρακτήρα. Πρέπει να υπογραμμίσω επίσης, κύριε Πρόεδρε, ότι η πρόταση αυτή έχει μπλοκαριστεί από το, από το Συμβούλιο. Από την Πολωνία που προεδρεύει αυτή τη στιγμή και από το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν αντίθετη θέση από αυτή με την Κομισιόν. Εν τέλει, η αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει την ε, αύξηση των ε, φορολογιών στην ενέργεια με το να αυξήσει την ε, φορολογία της εργασίας. Επομένως, αυτό κάνει κάτι στο οποίο δεν είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τη φορολογία της εργασίας. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι η μεθοδολογία της Κομισιόν για την αξιολόγηση αυτής της πρότασης μας φαίνεται πάρα πολύ αφισβητήσιμη. Αυτά. Thank you, Ayala Sender. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι έχουμε απλώς μια γνωμοδότηση για τα θέματα μεταφορών σε ένα ευρύτερο χώρο, ένα χώρο στον οποίο η Κομισιόν με κάποιους αξιόπαινους στόχους προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό φυσικά είναι ένα ερωτηματικό. Αν αντιμετωπίζει τις ε, εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο, δεν λαμβάνει υπόψη άλλα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά στην αγορά των καυσίμων και αν μπορούν να προκύψουν από εκεί άλλα προβλήματα πιο σοβαρά και επομένω θέτοντα σε μειονεκτική θέση το ντίζελ μπορεί να ευνοήσει άλλα καύσιμα τα οποία είναι ε, πιο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Επομένως και, και εδώ είναι θετικά τα κίνητρα που δίνονται αλλά σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι διευρυμένη είναι πολύ υψηλό το κόστος της ε, μετακίνησης των προϊόντων και της επιμελητίας και δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη να παραγνωρίσετε και το θέμα της, ε, του κόστους εργασίας. το κόστος μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις είναι αυτό το οποίο πλήττει ιδιαίτερα τις χώρες αυτές οι οποίες προσπαθούν να προσεγγίσουν τον πυρήνα της Ευρώπης και να ξεπεράσουν την περιφερικότητά του. Συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν εργαστεί πάρα πολύ στα θέματα των δικτύων και υπήρξαν κάποιες ε, ε, δηλώσεις της Επιτροπής μας και μας κυνηγάνε οι δημοσιογράφοι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η γνωμοδότηση αυτή που έχουμε και σέβομαι τις θέσεις που διατυπώθηκαν προηγουμένως ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να μετακινηθούμε προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτή η οδός που μας δίνει αυτό το νομοθέτημα. Πιστεύω πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί ώστε μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Μεταφορών να μην οξύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση κρίσης που αντιμετωπίζουν πολλά από τα κρατημέλη μας και πολλοί από τους τομείς δραστηριότητας και να μπορούμε να έχουμε και μια δυνατότητα πρωτοβουλίας στην ε, Ισπανία, παραδείγματος χάρη, γίνονται πρωτοβουλίες όπως τα ταξί γίνονται ε, υβριδικά. Και αυτή τη στιγμή ο κόσμος προσπαθεί να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει ακόμα ε, μια λίστα αναμονής για να περάσουν στο φυσικό αέριο σε υβριδική μορφή. Εμείς θα καταθέσουμε λοιπόν τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή για να μπούμε στην ουσία του θέματος. Είδα κάποιες από τις τροπολογίες της εισηγήτριας η οποία ασχολείται με θέματα τα οποία είναι ίσως λεπτομεριακά, όπως είναι η αθλητική ναυτική δραστηριότητα ή αυτά που λέει ο κύριος ε, Κράμερ, που ζητά να γίνουν αλλαγές οι οποίες μπορούν να γίνουν μοναχά σε διεθνές επίπεδο. Αυτά για μένα είναι δευτερεύοντα όμως. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την εισηγήτρια για όλα αυτά που έχει κάνει και φυσικά θα καταθέσουμε τροπολογίες για να συμπληρώσουμε αυτή την πρόταση η οποία από την πλευρά της Κομισιόν νομίζω ότι είχε σε στόχο να, να ταράξει τα νερά αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι δίνει καλές ειδήσει στον τομέα των μεταφορών. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να εξηγήσω ότι στόχο τη πρόταση είναι να υποστηρίξουμε την πολιτική για τι κλιματικέ αλλαγέ και την ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προσαρμόζοντα το εφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για την ενεργειακά προϊόντα και κάνοντά το να συνάδει με τι πολιτικέ αυτέ. Να ευχαριστήσω τη συντάκτρια γνωμοδότηση για την ε, γενικά θετική γνωμοδότηση που ε, συνέταξη ως προς την πρόταση αυτή, να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα. Όντως, στην πρόταση αυτή θέλουμε να εφαρμόσουμε το σύστημα αυτό τόσο στις θαλάσσιες όσο και στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Να αναφερθώ επίσης σε κάτι το οποίο ανέφεραν πολλά μέλη της Επιτροπής. Η πρόταση δεν ασχολείται με τη φορολογία των καυσίμων στο θαλάσσιο τομέα και στον τομέα της αεροναυτιλίας. Η πρόταση ασχολείται με το εφιστάμενο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει πλήρη εξαίρεση για την προμήθεια καυσίμων για την χρήση αυτή. Πιστεύουμε ότι επί του παρόντος δεν έχει έρθει ακόμα το πλήρωμα του χρόνου προκειμένου να γίνει μια σχετική πρόταση για πλήρη φορολόγηση των καυσίμων αυτών ούτε έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου προκειμένου να πούμε στα κράτη-μέλη ότι μπορείτε να το κάνετε εσείς μονομερός. Έχει γίνει μία ανάλυση στο παρελθόν, έχω αναφερθεί σε αυτό, η οποία έδειξε ότι η μονομερής δράση από τα κράτη-μέλη ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα είχε κάποια σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση όσον αφορά την μείωση των εκπομπών. Ανταυτού θα είχε πολύ επιζήμια επίπτωση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων μεταφορών σε σχέση με ανταγωνιστέ εκτό ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ θα υπήρχαν υποχρεώσει για αυτού, αλλά όχι για του ανταγωνιστέ από τι τρίτε χώρε. Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το ζήτημα αυτό, προτού προτείνουμε τέτοια φορολόγηση. Και γι' αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να προτείνει, μάλλον θα προτείνει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, αφού αρχίσει να ισχύει το πλαίσιο αυτό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και το διεθνέ πλαίσιο τη διεθνή συγκύρια και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. γίνονται κάποιες ε, προσπάθειες. Ε, διάβασα και ένα άρθρο σε σχέση με την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσον αφορά το ζήτημα αυτό και κάποιες συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια της Σύμβασης του Σικάγο για τις ε, αερομεταφορές. Συζητήσεις επίσης γίνονται και στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ακριβώς επειδή γίνονται παράλληλες συζητήσεις χωρίς να έχουν καταλήξει κάπου σε πολλά, διεθνά, σε πολλά άλλα διεθνή φόρα, θεωρήσαμε και εμείς ότι δεν είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε σχετική πρόταση. Να απαντήσω τώρα σε κάποιες άλλες παρατηρήσεις που γίνανε. Ο κύριος Κάνσκια νομίζω είπε ότι ε, θα γίνουν κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αυξήσεις στους δασμούς για τα αυτοκίνητα μέχρι το 2018 το 2023 μόνο θα δούμε επιπτώσει από την πρόταση αυτή, όταν θα υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να φορολογήσουν όλα τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται για τι μεταφορέ, χρησιμοποιώντα το ίδιο φορολογικό καθεστώ, τον ίδιο φορολογικό συντελεστή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μέχρι το 2023 τα κράτη-μέλη έχουν περίπου 12 χρόνια για να προσαρμόσουν το φορολογικό του σύστημα. Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή σε όλε τι παρατηρήσει που γίνανε. Πάντω, δύο μέλη αναφέρθηκαν στι ε, επιπτώσει που θα έχουμε στι ε, πιο απομακρυσμένες περιφέρειες Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πληγούν περισσότερο από άλλε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω τη πρόταση, αυτή πρέπει να σα πω τα κράτη-μέλη διατηρούν ένα μεγάλο βαθμό ευελιξία στο να καθορίσουν τελικά το επίπεδο φορολόγηση. Επομένω και ο περιφερειακό αυτό χαρακτήρα έχει ληφθεί υπόψη στην πρόταση που κάναμε για την θέσπιση των φορολογικών συντελεστών. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδες συγητέ και την Κομισιόν για τις παρατηρήσεις τους. Νομίζω ότι όλες οι επίτροπε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ασχοληθούν και με τα θέματα της αντιμετώπισης των κλιματικών στόχων και επομένως θα πρέπει στην νομοθεσία που εγκρίνουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορεί λοιπόν να χρηματοδοτείται στο διηνεκές ο αεροπορικός κλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΤΟΥΙ και οι άλλοι tour operators να αλωνίζουν με φτηνές πτήσεις στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι όπως είπε και ο κύριος Κράμερ έχει πράγματι δίκιο ότι τα πλοία στην ανοιχτή θάλασσα είναι πραγματική, πραγματικές εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων. Οι οργανώσεις ε, της, ε, οι οργανώσεις περιβάλλοντος στρέφονται τώρα κατά των κρουαζιεροπλοίων τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρώπη γιατί η μαζική αυτή κίνηση ουσιαστικά γίνεται πηγή και προβλημάτων. Τώρα ο κόσμος από την κατάσταση, από την ε, πορεία του ανέμου μπορεί να καταλάβει πόσα, πόσοι ρήποι έρχονται από το θείο και από τα καύσιμα που προχώνται από αυτά τα μεγάλα πλοία τα οποία κυκλοφορούν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια μεταφορά των μεταφορών στα, στους σιδηροδρόμους, αλλά αυτό πρέπει να γίνει και με κατάλληλη αναδιάταξη της φορολογίας. Αυτό είναι προϋπόθεση για να γίνει κάτι τέτοιο. Και δεν είναι ο μόνος συντελεστής που πρέπει να ληφθεί υπόψη για να λυθούμε το πρόβλημα. Δεν φτάνει μόνο η φορολογία. Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει στην Ευρώπη να ξεκινήσουμε με μερικά νέα συστήματα, όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών, κάτι το οποίο το κόμμα μου δεν θεωρεί ιδιαίτερα επιτυχές, αλλά τουλάχιστον έχουμε καταλήξει στο να υπάρχει ένα παγκόσμιο εμπόριο ε, εμπορίας για τα, για τα δικαιώματα εκπομπής που έχει οδηγήσει και σε κάποιους μηχανισμούς εφαρμογής που προστατεύουν το περιβάλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για την πρόταση της Κομισιόν και η γνωμοδότησή μας θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το πρώτο γύρο συζητήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ίσως είναι πρόωρο να μιλήσουμε για ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Μπορεί να, κάνουμε, να χρειαστεί να κάνουμε και κάποιους ακροβατισμούς για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. πει περιπτώσει προθεσμία τροπολογιών 21 Οκτωβρίου στι 12 η ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών 22 Νοεμβρίου και στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων 24 Ιανουαρίου. Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Έχετε κάποιο άλλο θέμα, διάφορο που θέλετε να θίξετε. Εάν όχι, η επόμενη συνεδρίασή μας είναι η 5η 10 Νοεμβρίου στις 9 η ώρα και ακολουθεί η 5η 21 Νοεμβρίου στις 3 η ώρα. Και κλείνει η συνεδρίαση. Ευχαριστώ όλους για την εργασία τους και τους διερμηνείς.